Um, colleagues, given that the... Συνάδελφοι, καθώς λέει ο Πρόεδρος και είμαι και η συγγήτρια για το πρώτο σημείο της Μερσίας Διάταξης, να τολμήσω να προτείνω να ξεκινήσουμε. Συμφωνούμε όλοι. Ομόφωνα, πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε επιτέλους στο σημείο ψηφοφορίας για τη συμφωνία με την Αυστραλία σε σχέση με τη διαβίβαση των PNR και τους καταλόγους ονομάτων επιβατών. Όσοι είναι παρόντες, δεν ε, νομίζω ότι χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσει. Ε, θα βρείτε ενώπιον σας ένα σύντομο κείμενο μιας ε, ενός σχεδίου σύστασης ε, και ένα σχεδίο μνημονίου κατανόησης νομίζω επίσης ε, κυκλοφόρησε χθε το βράδυ. Ξέρω ότι δεν είχατε πάρα πολύ χρόνο να το εξετάσετε, αλλά μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Και καθώς έχουμε πιέσει και τα άλλα όργανα να εργαστούν γρηγορότερα, ελπίζω να μπορούν να το δεχτούν όλοι, σε ό,τι αφορά στο χρονοδιάγραμμα. Προτείνω να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων σήμερα και να ψηφίσουμε το σχέδιο σύσταση στις 17 Οκτωβρίου και στη συνέχεια να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια στα τέλη του μήνα. Λοιπόν, η σύσταση, το σχέδιο σύσταση είναι πολύ σύντομο, αλλά υπάρχουν δύο δυνατότητες. Μπορούμε να συνενέσουμε ή να μην συνενέσουμε ακόμη. Εγώ θα πρότεινα να συνενέσουμε, να δώσουμε τη συγκαταθεσή μας, ε, όμως ε, για το επεξηγηματικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφερθούμε περαιτέρω μαζί με τους κοιόδης των άλλων ομάδων. Θέλω να αναφέρω κάποιες ε, σε ανησυχίες, γιατί από τη μία είναι αλήθεια ότι κατορθώσαμε να βελτιώσουμε τις προηγούμενες συμφωνίες, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ορισμό του σκοπού, έχει γίνει πιο αυστηρός, συνήθιζε να είναι πολύ ευρύ στα PNR, τα δεδομένα PNR χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό τώρα, περιορίζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για το σοβαρό διεθνές έγκλημα. Αυτό αποτελεί σαφή πρόοδο, αλλά υπάρχουν και κάποια θέματα όπου δεν έχουμε σημείωση επιτυχία ή πρέπει να δούμε κάποια πράγματα αν θα βγουν στην πράξη όπως ελπίζαμε. Κάτι που δεν πετύχαμε και αυτό θα είναι σχετικό και με μελλοντικές συμφωνίες PNR είναι μια κατάλληλη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Εδώ και χρόνια ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ε, δώσει ένα τέτοιο τεστ αναγκαιότητας και αναλογικότητας. Ε, έχουμε αρκετές τυχαίες περιστασιακές αποδείξεις, αλλά δεν έχουμε πραγματική απόδειξη της αναγκαιότητας και αναλογικότητας ε, ε, αυτής της ε, αδιάκριτης αποθήκευσης τόσων δεδομένων. Ναι, είναι χρήσιμα τα δεδομένα, δεν το αρνούμαστε. Είχαμε και τις επισκέψεις ε, ε επί που είχαμε την ενημέρωση από την Κομισιόν, ξέρουμε ότι μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα τα δεδομένα και απαραίτητα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν μου έχει αποδειχθεί ακόμη, γιατί πρέπει να αποθηκεύονται δεδομένα εκατομμυρίων αθών ανθρώπων για τόσο πολύ καιρό. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το επιλύσουμε για μελλοντικέ συμφωνίες. Και ένα άλλο σημείο ε, που διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θέμα της νομικής βάσης. Ξεκολουθούν να πεπισμένοι το άρθρο 16 της συνθήκης για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί τη νομική βάση και όχι τα δύο αντίστοιχα άρθρα για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Αν δείτε το ιστορικό των συμφωνιών PNR είναι προφανές το γιατί. Η αρχική συμφωνία PNR με τις ΗΠΑ υπεγράφει γιατί οι ΠΑΣ συνέλεγαν δεδομένα PNR. Τώρα, οι αερομεταφορεί ε, δυνάμει τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν επιτρεπόταν να δίνουν αυτά τα δεδομένα. Έτσι, λοιπόν, παρέβαιναν ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και για να διασφαλίσουμε ότι η διαβίωση των δεδομένων ε, σεβόταν τα πρότυπα προστασία των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνήθεια αρχική συμφωνία με τους Αμερικανούς. Έτσι λοιπόν είναι προφανές ότι ο στόχος τέτοιων συμφωνιών είναι η προστασία των δεδομένων και γίνεται ακόμη πιο προφανές ε, αν συνειδητοποιήσετε ότι δεν μιλάμε εδώ για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, γιατί μιλάμε για μονομερείς κυρίαρχες αποφάσεις ε, άλλων χωρών, τρίτων χωρών να συλλέγουν τέτοια δεδομένα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για αυτές τις χώρες ότι δεν μπορούν να συλλέγουν αυτά τα δεδομένα. Δεν θα το αποφασίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται για ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, αυτή είναι μια μάχη που χάσαμε, τουλάχιστον προς το παρόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει το άρθρο 60 να μην είναι νομική βάση, ούτε καν μερική νομική βάση, δεν γίνεται καμία μνήα σε αυτό. Μόνο μια πολύ αόριστη αναφορά που δεν έχει νομικό βάρος και νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό και Κάτι ακόμη που θέλω να πω για τις περιόδους αποθήκευσης. ότι τώρα να αποθηκεύονται το δεδομένα 5,5 έτη και, και ένα μέρος ε, αυτού του χρονικού διαστήματος ε, σε ανώνυμη μορφή. Τώρα τα 5,5 χρόνια μπορεί να είναι λογικό, μπορεί και όχι, αλλά δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, ούτε αιτιολογία. Από ό,τι φαίνεται επιλέγεται τυχαία Μέχρι πέρσι οι Αυστραλοί δεν αποδίκευαν τα δεδομένα, δεν βλέπω τι άλλαξε δηλαδή μεταξύ του 2010 και τώρα. Αλλά για να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα θα εξακολουθούσα να συνιστώ να συγκατατηθούμε σε αυτή τη συμφωνία, όχι γιατί είμαστε 100% ικανοποιημένοι με αυτή, όχι γιατί δεν υπάρχουν ανησυχίε που παραμένουν, αλλά δείτε όλες τις επιλογές που έχουμε. Νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή είναι να συνενέσουμε γιατί αν δεν συνενέσουμε θα συνεχίζουν να διαβιβάζονται τα δεδομένα εκτός και να αποφασίσουμε να διακόψουμε κάθε ενέργεια κυκλοφορία, δεν φαίνεται βέβαια αυτό να είναι και πολύ ρεαλιστικό. Θα συνεχίζονται λοιπόν να, να διαβιβάζονται τα δεδομένα και νομίζω ότι έχουμε εδώ επιτάπητος είναι μια αποδεκτή συμφωνία. Δεν είναι ένα καλό επίπεδο προστασίας, ε, ακόμη και με όλες τις παρεκκλήσεις που μόλις σας ανέφερα. Αυτό σας συστήνω λοιπόν εγώ. Okay, thank you, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Ινβέλτ για την παρουσίαση του σχεδίου συστάσεως για να συνενέσουμε στη Συμφωνία Αυστραλίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τα PNR και τώρα θα ακούστε τον ε, κύριο Βος ε, και ίσως πριν όμως μιλήσουν οι ευρωβουλευτές ε, θα έπρεπε να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν όμως από αυτόν τον κύριο Βος. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για την ε, συνόψιση των ε, απόψεών μας διότι νομίζω τα παρουσιάστε πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι αν κοιτάξουμε ε, τον στόχο του εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε μεγαλύτερη προστασία δεδομένων ή περισσότερη προστασία δεδομένων πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι σε όλα τα σημεία αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουμε επιτύχει το στόχο μας, ιδίως διότι θα, είχαν, θα υπήρχαν επιπτώσεις αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο δεν αναλάμβανε αυτή την πρωτοβουλία και θα υπήρχαν μόνο μειονεκτήματα στις εξελίξεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό και ενδεχομένως θα είχαμε τελείως άλλες μορφές ε, αεροδρομίων ή άλλα προβλήματα σχετικά με τα δεδομένα ε, και την προστασία τους. Γι' αυτό και έχω το συνέστημα ότι όσο μπορέσαμε να κρατήσουμε τον έλεγχο και κατά κάποιον τρόπο να εφαρμόσουμε το σύστημα αυτό, ε, είτε πρόκειται για διημερή συμφωνία είτε για ανταλλαγή με τις αεροπορικές εταιρείε, δεν υπάρχουν πολύ καλύτερες λύσεις που θα μπορούσαν να ισχύσουν και γι' αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και θα πρέπει να συνενέσουμε παρόλο που όπως είπα υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είμαστε σε καλύτερη μοίρα αλλά όσον αφορά τις επιπτώσεις και τα ενάψματα προς τις Ηνωμένε Πολιτείες θεωρώ ότι το σύστημα αυτό είναι καλό και θα πρέπει να το στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Και τώρα ε, οι σκιώδεις εισηγητές, η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, θέλω να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα και να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον ενθουσιασμό της διότι μας έχει πει και στο παρελθόν όπως και τώρα ότι κανείς από μας ε, δεν είναι ίσως ικανοποιημένος 100% με την πρόταση που εξετάζουμε αλλά συνήθως σπανίως καταλήγει καταλήγουμε σε συμφωνίες ή σε οδηγίες που ικανοποιούν τους πάντες γιατί και εδώ χρειάζεται στο Κοινοβούλιο να καταλήγουμε σε συμβιβαστικές λύσεις διότι χωρίς μία συμφωνία οι αεροπορικές εταιρείες ε, δεν ε, θα μετέδιδαν ανεξέλεγκτα τα στοιχεία και πιστεύω ότι αν πρόκειται ε, για διμερείς συμφωνήσεις αντί για μία ενιαία κάλυψη και συμφωνία εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως οι περισσότερες διατάξεις θα ήταν μενέστερες. Γι' αυτό και συμφωνώ να υπάρχει ε, τέτοιου είδους συμφωνία διότι δεν μπορούμε ε, να απαγορεύσουμε σε κανένα κράτος να προστατεύσει τα εξωτερικά του σύνορα και θα μπορέσουν βέβαια περαιτέρω αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιηθούν και για άλλους στόχους. Δεν μπορούμε αυτό να το αλλά εδώ πρέπει να ισχύσουν ορισμένες προϋποθέσεις προστασίας και γι' αυτό όπως σας είπα μπορεί να μην είμαι ικανοποιημένη 100% αλλά είναι ε, καλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και γι' αυτό νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ορισμένες κριτικές προτάσεις μπορεί ε, να ε, αποδεχτεί αυτό το, το θέμα. Τώρα ο κύριος Κίρκοπ έχει το λόγο. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα σήμερα το πρωί. Κάτι σύντομο θέλω να πω. Θέλω να ευχαριστήσω την αδελφή για τη δουλειά της για το θέμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και θέλω να τονίσω και από τη δική μου σκοπιά πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα ε, που θα προστατεύονται ορθώς και σίγουρα υπάρχουν πολλές βελτιώσεις εδώ, κυρίως ό,τι αφορά την αποθήκευση των δεδομένων. Νομίζω ότι σημειώσαμε πραγματική πρόοδο και πιστεύω προφανώς ότι είναι καιρός για μας ε, να είμαστε υπευθύνοι και να συνενέσουμε Μπορεί να μην είμαι 100% αλλά είμαι 95,3% ικανοποιημένο. Ε, και παρά την αλλαγή στην μερική διάταξη είμαστε γνωρίζουμε όλοι ότι θα διαβάσει το δεδομένο εξάρτητα από τις συμφωνίες που θα υπογραφούν ε, αυτή την ε, πραγματικότητα τη γνωρίσαμε πρόσφατα, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να έχουμε αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον να ρυθμίζουμε και να προστατεύουμε τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών και νομίζω ότι αποτελεί πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με ότι είχαμε νωρίτερα. Έτσι λοιπόν, συγχαρητήρια και φυσικά θα υπάρχει πλήρη υποστήριξη από τη δική μου ομάδα. Uh, Ο κύριος Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί πρέπει να φύγω για μια άλλη επιτροπή, θα έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Ε, είδατε φτάσει και κάποιο συνάδελφο με τον οποίο συμμεριζόμαστε τι ίδιε Ε, Εδώ θέλω να σας πω ότι γνωρίζω ότι η συμφωνία είναι καλύτερη σε σχέση με αυτή που έχουμε με του Αμερικανού. Ξέρω ότι η ροή των δεδομένων δεν θα σταματήσει, αλλά με ανησυχεί ο χρόνος της αποθήκευσης. Όπως ε, ξέρουμε δεν ε, υπάρχουν σαφή πρότυπα για το χρόνο της αποθήκευσης, αλλά Νομίζω ότι πρέπει να ανησυχούμε για τη συνέπεια των ίδιων των δεδομένων μα, ε, όταν χρησιμοποιούμε την ομολογία εντό τη Ευρώπη, ε, για να λέμε ότι πρέπει να αποθηκεύονται τα δεδομένα για κάποιου μήνε, όχι για χρόνια. Τα 5,5 χρόνια είναι πάρα πολύ. Επίση, ανησυχώ για την πρόθεση των δεδομένων σε τρίτε χώρε, αλλά καθώ πρέπει να φύγω θα σταματήσω εδώ και ίσω ε, μπορεί να παρουσιάσει κάποιε από τι κοινέ ανησυχίε μα. Thank you then. Μάλιστα. Αν ο κύριος Άλμπρεχτ θέλει να ακολουθήσει τον κύριο Ταβάρης, θα ήθελα να μιλήσω για τη συμφωνία, αλλά αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής του μέσης διάταξης για μένα είναι τελείως απαράδεκτη. Δεν μου επιτρέπει να εργαστώ όπως θέλω. Πήρα το ηλεκτρονικό μήνυμα, μήνυμα χθες το βράδυ, δεν προλαβαίνω. Δεν μπορούμε να εργαζόμαστε έτσι. Εγώ δεν μπορώ με αυτόν τον τρόπο. Για δε τη συμφωνία υπήρχαν πολλά, υπήρξαν πολλά ψηφίσματα για το PNR. Είχαμε πει ποιες είναι οι αρχές που δεχόμαστε και συγκρίνοντας τη συμφωνία με τα ψηφίσματα αυτά μεταξύ Αυστραλίας και Ένωσης για το PNR. Δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε αυτά που είχαμε ζητήσει, ιδιαίτερα τις προτεραιότητές μας. Το θέμα του profiling δεν αναφέρεται καν, ενώ για μας ήταν πάντοτε για όλο το Κοινοβούλιο σημαντικό θέμα. Ζητήσαμε να μην συμπεριλαμβάνεται profiling. Και τουλάχιστον ζητούσαμε να υπάρχει σαφής ορισμός του τι εννοεί. Δεν νομίζω λοιπόν ότι τέτοιο μέτρο θα γίνει δεκτό από το Κοινοβούλιο. Έτσι δημιουργείται προηγούμενο και για άλλες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. και για τα μέτρα που θα λάβουν οι χώρες μέλη. Υπήρξαν πολλές προσφυγές σε συνταγματικά δικαστήρια για θέματα κρατήσεων χωρίς δικαιολόγηση και δεν νομίζω ότι πρέπει να το εγκρίνουμε. Κύριε Άλμπεριχ, όλοι σεβόμαστε αυτά που είπατε και τα εκτιμούμε ιδιαιτέρως και δεόντως, αλλά αλλά λέγω, για να απαντήσω στο πρώτο σας σχόλιο για τον τρόπο εργασίας της Επιτροπής ΕΛΕΦ, εδώ είμαστε πάνω από 50 και κανένας, ούτε καν εγώ, δεν υπάρχει που να μην έχει και άλλες ανηλυμένες πολιτικές υποχρεώσεις. Μα γι' αυτό έχουμε ημερήσια διάταξη, λέει ο κύριος Άλμπρεχτ. Ναι, αλλά καμιά φορά, επειδή έχουμε υπερφορτωμένη ημερήσια διάταξη και φόρτο εργασίας, κάποτε μπορεί να συμβεί ότι κάποιος, όπως έγινε χθες με την κυρία Ιντφελντ, να ζητήσει μεταφορά της σειράς ορισμένων σημείων της ημερήσιας διάταξης. Έχει δικαίωμα να ζητήσει να είναι το πρώτο θέμα, ας πούμε, όπως ζήτησε για σήμερα. Και αποφασίσαμε να το δεχτούμε, συμφωνήσαμε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι αρνητικό και ότι μπορούμε να λέμε ότι είναι απαράδεκτες καταστάσεις και τέτοια πράγματα. Ήταν λογικό το αίτημα, συμφωνήσαμε να δεχτούμε αυτό που ζήτησε η κυρία Ίνφελντ χθες και το θέμα ε, δεν είναι κάτι που γίνεται συνεχώς, είναι εξαιρετικό. Και γι' αυτό βρίσκω το αίτημα φυσικό και λογικό να παραμένουμε ελαστικοί σε τέτοιου είδους αιτήματα για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως εξελίσσονται. Φαντάζομαι ότι αυτή την εξήγηση μπορείτε και εσείς να τη δεχτείτε. Τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Μπρόνς και μετά και μετά θα μας ενημερώσει η Κομισιόν ε, και θα ακούσουμε και τον κύριο Ίνβελτ. Ναι, ε, Συγγνώμη, δεν εμφανίστηκα στην ώρα μου και δεν έχω καμία δικαιολογία. Δηλαδή, μπορεί να απαντήσατε ήδη στην αρχική σα εξήγηση, αλλά είπατε ότι ακόμη και αν δεν υπογράφαμε τη συμφωνία, ούτω ή άλλω θα διαβάζονταν και θα αποθηκεύονταν τα δεδομένα. Αυτό λοιπόν πρέπει να σημαίνει ότι οι πληροφορίε που συμπεριλαμβάνουν είναι αυτές που χορηγούνται σε συνηθισμένη βάση, όπως παραδείγματο χάρη και λεπτομέρειες πιστοτικής κάρτας και θα επεκτείνονταν σε πληροφορίες που, στην, που δίνονται στην κυβέρνηση σε σχέση με τις αιτήσει για θεώρηση. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι απαντήσατε λοιπόν την ερώτησή μου. Κύριε Thank Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σοφή για την εισαγωγή της ε, σήμερα. Ακόμη και εγώ δεν είμαι σκιώδη για την ομάδα μου. Ε, λείπει η σε την ομάδα μου, ζήτησε να διαβάσω πέντε σημεία. Το πρώτο σημείο έχει ως εξή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύο περιπτώσεις, στις 5 Μαΐου 2010, και στις 11 Νοεμβρίου 2010 υιοθέτησε ψηφίσματα σχετικά με απαιτήσει για μια συμφωνία PNR ώστε να είναι αναλογική. Κάποιες ε, σημαντικές απαιτήσει δεν ε, υπάρχουν στη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε τα δεδομένα PNR μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο για να καταπολεμηθούν η τρομοκρατία σύμφωνα με την απόφαση πλαίσιο 2002-475 ε, αλλά έχει μεγαλύτερο ε, πεδίο εφαρμογή οδηγία θα χρησιμοποιηθεί και για να καταβληθεί το σοβαρό διεθνέ έγκλημα. Ε, δηλαδή οτιδήποτε τιμωρείται στην Αυστραλία με μέγιστη ποινή τουλάχιστον 4 χρόνια και εν μέρη έχει εφαρμοστεί στο εξωτερικό αυτό καλύπτει πάρα πολλά αδικήματα και πολλά που δεν θεωρούνται σοβαρά ή τρομοκρατικά αδικήματα. Δεν υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες για να επιτραπεί ε, η μεταφορά των δεδομένων σε τρίτες χώρες όπως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβει τα δεδομένα μια τρίτη τη χώρα. Απλώ το μόνο που πρέπει να κάνει είναι ότι θα σεβαστεί τι εγγύσει όπω ορίζονται στη συμφωνία. Όμω δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει ακόμα αποδείξει ότι το PNR είναι αναλογικά και όπως συζητήθηκε Επίσης, η απόδειξη για τη διατήρηση των δεδομένων PNR για 5,5 χρόνια είναι κάτι απαραίτητο και εξακολουθεί να λείπει αναλογικότητα. Μετά από τρία χρόνια θα καταστούν ανώνυμα τα δεδομένα και θα αποκοιτεύονται για ακόμη 2,5 χρόνια. Αυτό, ενώ ακούγεται καλό, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί γίνεται σαφές από το κείμενο ότι μετά από την ανωνυμοποίηση μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα για ορισμένες έρευνε αν χρειαστεί. Έτσι λοιπόν, τίποτα ουσιαστικό δεν έχουμε εδώ που θα καθιστούσε πραγματικά πραγματικά ανώνυμα δεδομένα, αλλά έχουμε κάποια ε, δεδομένα ε, και καλυμμένα για τα οποία δεν ε, είναι δύσκολη πρόσβαση. Έτσι λοιπόν 5,5 χρόνια αποθηκεύονται τα δεδομένα και όχι τρία και από το Αυστριαλενό Ίδρυμα για την εμπιστευτικότητα μας είπαν ότι τα πρότυπα της Αυστραλίας είναι πολύ χαμηλότερα από τις Ευρωπαϊκές Ένωσες, γι' αυτό ποτέ η Αυστραλία δεν έχει λάβει την κατάλληλη βαθμολογία. Αυτά είναι τα σχολεία της συναδέλφου. Ευχαριστώ κύριε Βερζάτ. Ναι κύριε Πρόεδρε, θα συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος Τριανταφυλλίδης. Συμφωνώ με αυτά που λέγονται και ιδίως από τους συναδέλφους Σταβάρες και Άλμπρεχτ. Βεβαίως ε, δεν είμαστε στην ίδια κατάσταση με την ε, ε, συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά εάν κατάλαβα καλά αυτά τα οποία είπε η Σόφη Ίνβελτε πρέπει να έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις για τις εξελίξεις και θέλω να αναφερθώ σε τέσσερα σημεία που συνάδουν με παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Ποιες είναι δηλαδή δηλαδή παραδείγματος χάρη οι σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, δηλαδή γιατί χρειάζονται ε, μέτρα για τον, ε, την τρομοκρατία. Πάντοτε θεωρήσαμε ότι χρειάζεται μη, ένας ακριβής ορισμός ε, των όρων και εδώ δεν έχουμε μία αναλογική αντιμετώπιση. Ποια στοιχεία μπορούν να μεταβιβάζουν και εκεί υπάρχει κάποια σάφια γιατί η διάρκεια της κατακρατήσεως των στοιχείων έχει αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία και γιατί να υπάρχει αυτή η υπερβολική ε, προθεσμία η οποία δεν ε, έχει καμία σχέση με το παρελθόν και τέλος ε, όσον αφορά τις, ε, ε, τα θέματα τα οποία οδηγούν σε συνεχείς διαφορές, τι συμβαίνει γιατί κανείς δεν μου εξήγησε. Πριν όμως ξαναδώσω το λόγο στον, στην κυρία Ινβέλτ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Νταλμέιντα. Ευχαριστώ. Νομίζουμε ότι η συμφωνία αυτή είναι πολύ ικανοποιητική, πρέπει να ικανοποιήσει το Κοινοβούλιο και συνάδει με τις ε, οδηγίες ε, του Συμβουλίου και νομίζουμε ότι σοσκελίζει την ασφάλεια ε, με την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία και νομίζω ότι έτσι θα απαντήσω στα περισσότερα ερωτήματα η ε, περίοδος κατακράτησης των στοιχείων ήταν η πλέον δύσκο το πιο δύσκολο θέμα διότι έχει παραμείνει στα 5,5 χρόνια και δεν έχει αυξηθεί. Αλλά η Αυστραλία ε, ζητά να έχει πρόσβαση σε όλα τα τα στοιχεία για τα πρώτα τρία χρόνια και μετά από τρία χρόνια τα στοιχεία που ε, ταυτοποιούν και εντοπίζουν τον επιβάτη θα αποκρύπτονται και αυτό θα ελεγχθεί και πάλι σε την κοινή εξέταση η οποία θα γίνει ένα χρόνο μετά την υπογραφή της συμφωνίας και θα δούμε εάν ε, αυτή η κατιούσα πρόσβαση ε, μετά τα 5,5 χρόνια έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά ή όχι. Θεωρούμε ότι όσον αφορά το στόχο έχουμε μια εξαιρετική ε, συμφωνία που καλύπτει πλήρως ε, τους λόγους για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν ε, τα PNR για να ερευνά κανείς και να διώκει το ε, ε, ε, τα σοβαρά εγκλήματα και ιδίω διασυνοριακά και ιδίω την τρομοκρατία και εφόσον συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών διεθνικών εγκλημάτων όταν δηλαδή ε, υπάρχει νομική ε, σαφήνεια ε, και καθορίζεται από ποινές πέραν των τεσσάρων ετών θα πρέπει όμως να συνάδει ε, με τις συμφωνίες ε, του ΟΗΕ σχετικά με τα διεθνή εγκλήματα και βλέπουμε στο άρθρο 20 ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να μεταφέρονται δια συγκεκριμένης μεθόδου και ε, υπάρχει συνεργασία για την ε, ε, για την δικαστική, στο δικαστικό τομέα με την Αυστραλία ε, και θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Europol και την Eurojust και θα πρέπει ε, να ε, κινείται μέσω αυτών των οργανισμών για να δοθούν πληροφορίες σχετικά με τα PNR στην ασφαλεία. Βεβαίως δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των ε, επιβατών να απαγορεύεται η μετάδοση των ευαισθητών στοιχείων και ε, όλα αυτά να καλύπτονται από τον Αυστραλό ε, Επίτροπο για τα θέματα της ασφαλείας να μην υπάρχουν ε, στοιχεία PNR τα οποία μπορούν να βλάψουν τους επιβάτες γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρχει καθορισμένο προφίλ το οποίο να οφείλεται σε αυτή τη συμφωνία του επιβάτη και να ε, έχουμε προβλέψει την επισκόπηση και την ε, διόρθωση των στοιχείων και ε, για τις ε, τρίτες χώρες θα πρέπει μεταφορές να ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και να λαμβάνονται υπόψη μόνο κατά περίπτωση. Επίσης οι υπεύθυνε αρχές των κρατών μελών πρέπει να ενημερώνονται ε, αν υπάρχουν στοιχεία ενός υπηκόου τους που με μεταδίδονται σε ένα τρίτο κράτος. Βέβαια είπαμε ότι θα υπάρξει μία αναθεώρηση μετά την υπογραφή και ε, θα ε, και ε, θα ε, μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ε, την εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Είχαμε ήδη δύο συνεδριάσεις επικοδομητικέ του θόμεατο με τους Ευρωβουλευτές και θα υπάρξουν κι άλλες εάν χρειαστούν. Ευχαριστώ κύριος Γκαζίνσκι εν ονόματι της Πολωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Θέλω να προσυπογράψω επί Κομισιόν, αλλά και ένα πολύ συγκεκριμένο τμήμα της συμφωνίας που συνήθει. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το δει κάποιος αμέσως όταν αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας, στο Συμβούλιο. Ακούγοντας επίσης και τις ιδιαίτερες θέσεις των μελών της Επιτροπής, ε, κατάλαβα ότι θα ήταν σοφό να οθήσει την Κομισιόν ως ένα συγκεκριμένο βαθμό και η Κομισιόν να ε, επέστρεψε στις διαπραγματεύσεις με τους Αυστραλούς και υπάρχει μια κοινή δήλωση που προσαρμοζόταν στο κείμενο της συμφωνίας. Δηλαδή, η δήλωση δεν αλλάζει τη φύση του κειμένου, αλλά τονίζει τρεις συγκεκριμένα στοιχεία. Ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός που αφορά το reporting θα συσταθεί και οτιδήποτε θα γίνει ε, οποιοδήποτε ε, μεταφορά δεδομένων θα σέβεται την αρχή της περίπτωση ανά περίπτωση. Και η διαβούλευση με την Αυστραλία θα είναι ένα από τα κύρια στοιχεία της διαδικασίας ε, που θα πηγάζει από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Αυτό υπογραμμίζει τη βούληση των Αυστραλών να μείνουν σε επαφή μαζί μας ε, και πρέπει να ευχαριστήσω εγώ ξανά με Προεδρία στην Ιδίω γιατί μπόρεσε κατά κάποιο τρόπο να ξανανοίξει τι διαπραγματεύσει και να κινηθεί έναντι των Αυστραλών. Και αυτοί τελικά συμφώνησαν. Βέβαια, αυτό δεν θα έχει γίνει ποτέ χωρί ε, και τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη βούληση των Αυστραλών να κατευθυνθούν προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάλιστα, κύριε Ιντβελτ, εσεί έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε κάπως γιαστικά και το ξέχασα. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης γιατί συνεργαστήκαμε και εργαστήκαμε ως ομάδα και φυσικά θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ως ομάδα γιατί έχουμε και άλλες συμφωνίες στο μέλλον. Λοιπόν, ε, καταρχήν ε, για τους Πρεσίνους και για την ΚΟΕ και για την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας πω ότι μην απατάστε, δεν είμαι 100% ικανοποιημένη. Ο κύριος ε, Νιουνιές ε, τοποθετήθηκε. Ναι, ε, υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία στη συμφωνία, αλλά ξέρετε ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή έχουμε τώρα ένα καλό νομικό ορισμό αλλά εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα για εξαιρέσει. Ξέρετε ότι ο Ευρωπαίος Αποπτής Προστασίας των Δεδομένων έχει εκφράσει ανησυχίες για το θέμα αυτό και αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο κείμενο αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τις επιλογές που έχουμε επιτάπητος. Υπάρχει δυνατότητα να επαναδιπραγματευτούμε το κείμενο της συμφωνίας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Η δυνατότητα είναι να πούμε ναι ή όχι σε σχέση με αυτό που έχουμε τάπητος. Αν υπήρχαν διάφορες επιλογές, εγώ αυτό θα προωθούσα ως εισηγήτρα, πιστέψτε με αλλά δυστυχώς ε, πρέπει να δούμε σε ποια πραγματικότητα ζούμε. Και το ερώτημα είναι, τελικά θα γκρίνουμε αυτή τη συμφωνία ή όχι. Επίση, σε σχέση με όσο υποθήκαν από γκο και πρασίνους να πω ότι συμφωνώ. Ε, Πολλέ από τι κυρίε ανησυχίε δεν υπάρχουν στο ίδιο το κείμενο της συμφωνίας, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο. Όπως είπα, η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα ακόμη δεν έχουν αποδειχθεί επαρκώς. Αλλά αυτό δεν αποτελεί τμήμα του κειμένου της συμφωνίας. Αυτό θα πρέπει να το έχει κάνει η Κομισιόν. Και αυτό πρέπει να κάνει για μελλοντικέ συμφωνίες και για το ευρωπαϊκό PNR. Και ένα άλλο θέμα είναι η νομική βάση. Αλλά φυσικά γι' αυτό δεν αποτελεί τμήμα της ίδιας της συμφωνίας. Αν δείτε τα δύο ψηφίσματα που υθετήσαμε, και στο οποίο αναφέρθηκα Μάιο και Νοέμβριο πέρσι, η συμφωνία σέβεται πολλά από τα κριτήρια που είχαμε συστήσει και έτσι λοιπόν πολλές από τις ανησυχίες βρίσκονται εκτός του διατακτικού. Για την κυρία Βερζιά κάτι να διορθώσω. Τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν είναι ορθώς προσδιορισμένα Πάντοτε γνωρίζουμε ποια δεδομένα μπορούν να συλλεφθούν και ποια όχι. Δεν υπήρχε ποτέ θέμα με αυτό. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες για το υπεραιτέρω διαβίβαση, τώρα περίοδο διατήρησης. 5,5 χρόνια φαίνεται να είναι μια τυχαία επιλογή, ίσως ε, να είναι σωστή, να είναι λανθασμένη. Αυτή η περίοδος να είναι πολύ μεγάλη, πολύ μικρή, δεν το ξέρουμε η Κομισιόν. Θα πρέπει να το έχει αποδείξει αυτό και πρέπει να το πράξει. Σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό των δεδομένων, το profiling, η συμφωνία δεν αναφέρει το profiling. Αυτό τώρα μπορεί να είναι καλά να και κακά ναι, δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι αποκλείεται ο χαρακτηρισμός, αλλά μπορεί να σημαίνει ότι επιτρέπεται. Και η Κομισιόν λέει ότι δεν ε, υπάρχουν αυτόματες αποφάσεις, αυτό δηλώνεται στη συμφωνία και επομένως δεν θα υπάρξει profiling, νομίζω ότι κάνετε λάθο, γιατί οι τι αποφάσει και το profiling, ο χαρακτηρισμός είναι πολύ διαφορετικά πράγματα και αν διαπραγματεύτηκε η Κομισιόν βάσει αυτή τη υπόθεση, λάθο κάνατε νομίζω. Δεν έχουμε εγγύηση ότι δεν θα υπάρχει profiling, έχουμε την εγγύηση ότι δεν θα υπάρχουν αποφάσει που θα λαμβάνεται αυτοματοποιημένα. Αυτό δεν είναι όμω το ίδιο. Και χαίρομαι που ακούω ότι προβλέπετε και είναι αναθεώρηση μέσα σε ένα έτος. Αυτό είναι κάτι θετικό. Σε σχέση με το περιορισμό του πεδίου εφαρμογή, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά, υπάρχουν πιθανέ εξαιρέσει. Παραδείγματο χάρη, αναφέρεται το θέμα τη δημόσια υγεία. Μα συγχωρείτε, η δημόσια υγεία δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατία ή με το σοβαρό διεθνέ έγκλημα. Α είμαστε ειλικρινεί. Θα συνιστούσα λοιπόν να υπερψηφίσουμε, αλλά δεν συστηνώ για να υιοθετήσουμε τον ίδιο τόνο που ακούσαμε μόλις ε, και τρία τελικά σχόλια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται όλα τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν ε, ή να συγκεντρωθούν στη συμφωνία αυτή. Ξέρουμε ότι θα υπάρχουν αποχές, τουλάχιστον ένα μεγάλο κρατισμένο θα πόσχει. Δεύτερο. Ο Πίτροπος έκανε μια δημόσια δήλωση στην Ολομέλεια, υπάρχει στα πρακτικά. Και θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό σε μια ανταλλαγή επιστολών. Η επίτροπο, με συγχωρείτε, η δεσμεύτηκε για να παρουσιάσει προτάσεις ε, για την αστολή ή ε, την καταγγελία της Συμφωνία. αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήσει από την Κομισιόν να πράξει κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι σαφέ στη συνθήκη για το ποια πρέπει να είναι η διαδικασία. Αλλά υπάρχει πολιτική συμφωνία και θέλουμε πριν πάμε σε ψηφοφορία να έχουμε μια επιβεβαίωση. Και τελευταίο σχόλιο, αυτό δεν αφορά τη συμφωνία με την Αυστραλία. Η Κομισιόν όμω πρέπει να κατανοήσει με σαφήνεια το εξή. Εμεί συζητήσαμε εδώ και πολλά χρόνια πολλά πράγματα και υπάρχουν πολλέ ερωτήσει που μένουν αναπάντητε. Όμως η Κομισιόν θα πρέπει να παράσχει το εξή πριν να σκεφτούμε να ψηφίσουμε μια συμφωνία με τι ΗΠΑ. Και αυτό είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει τι διμερέ συμφωνίε με τα κράτη-μέλη. Δύο έχουν συναυτεί τόσο πρόσφατα όσο φέτος το καλοκαίρι. Και έχουμε και εκεί αναφορέ στο PNR. Γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι διαπραγματευόμαστε, αν ταυτόχρονα πίσω από την πλάτη μα τα κράτη-μέλη επίση διαπραγματεύονται για τα PNR. Δεν έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει με την Αυστραλία, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το αποσαφενίσει η Κομισιόν και μάλιστα καταπηγόντως ε, και η απάντηση ότι δεν συνεργάζονται τα κράτη-μέλη δεν αρκεί. Θέλουμε αυτή τη διευκρίνηση. Αυτό έχω να πω. Συνάδελφοι, θα συνιστούσα να διαβάσετε το επεξηγηματικό σημείωμα. που Εκπονήσαμε συνεργασία με τους Σκιώδης, αλλά νομίζω ότι η επεξηγηματική δήλωση θα σας παρουσιάσει με μεγαλύτερες λεπτομέρειες ε, κάποιες από τις κυρίες ανησυχίες και τις προσδοκίες που έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Τώρα πρέπει να σας ανακοινώσω ότι οι διαδικαστικές τροπολογίες έχουν ως διορία 15 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Και η ψηφοφορία στην ΕΛΕΦ θα γίνει 17 Οκτωβρίου. 17 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε το, για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν όσους συμμετέσχουν στην συζήτηση αυτή και συνεχίζουμε με το επόμενο μας θέμα που αφορά την έκθεση του κυρίου Ντίαθ Ντεμέρα. την, ανα... την τροποποίηση του κανονισμού για τις θεωρήσεις. Πέρι του καταλόγου τρίτων χωρών υπήκοπη των οποίων προπόκειται στην υποχρέωση θεώρηση για την διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου των τρίτων χωρών υπήκοπη των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. είναι το θέμα των θετικών και αρνητικών καταλόγων θεωρήσεων και θα μας μιλήσει ο εισηγητής ο κύριος Δίας Δεμέρα και μετά θα μιλήσουν και άλλοι άμα θέλουν καθώς και η Κομισιόν και ο πρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας ο εισηγητής κύριος Δίας Δεμέρα Γκαρθία Κονσουέγρα Ευχαριστώ Πρόεδρε Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζουν, είχα την δυνατότητα να παρουσιάσω την εκθέση αυτή πριν ένα μήνα περίπου με την συνεργασία Συμβουλίου και Κομισιόν. Έτσι λοιπόν, αν θεωρήσω την είναι μου, αν το θεωρείτε την μου, μπορώ να αναφέρω και πάλι τα επιχειρήματα που είχα αναφέρει τότε, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο, κατά την άποψή μου, θα ήταν να ακούσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο σχετικά με τις εξελίξεις ε, του θέματος ε, στους κόλπους του Συμβουλίου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα κατάλληλα στοιχεία, τα κατάλληλες ε, πληροφορίες, να έχουμε επικαιροποίηση επί αυτής της διαδικασίας της διαπραγματευτικής όπου ξέρουμε ότι υπήρχαν και υπάρχουν ορισμένα στοιχεία αποκλήσεων. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και το Κοινομέι Βούλιο πρέπει να γνωρίσουν ε, τι ακριβώς, ε, πώς ακριβώς έχουν εξελίξει στο ιστορικό του Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν, να συμφωνείτε, Πρόεδρε, να δώσουμε τη δυνατότητα να τοποθετηθούν εκπρόσωποι Συμβουλίου και Κομισιόν και αν δεν το επιθυμούν, εγώ τότε θα παρουσιάσω και την έκθεση. Ευχαριστώ. Ας ακούσουμε τώρα τους Σκιώδης. Όχι. Να ξαναπώ. Είπα ότι θα ε, ήταν καλό να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο Συμβούλιο. Να δώσουμε το λόγο στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν. Με συγχωρείτε, εγώ μιλούσα όταν κάνατε αυτή την πρόταση. Βεβαίως, σας κατανοούμε. Έτσι λοιπόν, να ακούσουμε καταρχήν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πάλμαν ή τον κύριο Καρσία Μαρτίνες, πρόσωπος Κομισιόν. Θέλετε εσείς πρώτο λόγο ή το Συμβούλιο. My colleague Mr. Palman is ο συνάδελφός μου κύριος Πάλμεν θα έρθει σε λίγο, γι' αυτό παρακαλώ πρώτα την Πολωνική Προεδρία να μιλήσει. Ωραία, η Πολωνική Προεδρία, ο κύριος Γιαζίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ παρακολουθώ και το θέμα του PNR και τις θεωρήσεις. Θα ήθελα να σας δώσω μία σύντομη πληροφόρηση Φαντάζομαι ότι μπορώ ως προς αυτό να μιλήσω και για τα δύο όργανα Κομισιόν και Συμβούλιο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει πολλές αντιρρήσεις στα κράτη-μέλη ως προς την πρόταση της Κομισιόν και αυτό είναι θετικό. Με την εξαίρεση ενός δύο θεμάτων που θα αναφέρω τώρα, η πρόταση ως έχει θεωρείται ως καθαρά τεχνική. Βέβαια, το θέμα της συνεργασίας με την Τουρκία ή το θέμα της προσωρινής επαναφοράς των θεωρήσεων ε, δημιουργεί πολιτικές διαμάχες και αυτό είναι κατανοητό. Απαρόλα αυτά νομίζουμε ότι μπορεί να λυθεί εύκολα επί της Πολωνικής Προεδρίας. Το πρώτο θέμα που θέλω να θίξω αφορά το θέμα της αμοιβαιότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έγινε σεβαστή η αρχή της αμοιβαιότητας. Αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στην Κομισιόν και θεωρούμε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να λύσει και αυτά τα εναπομείναντα προβλήματα. Ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό αφορά την Τουρκία. Η πρόταση της Προεδρίας εδώ είναι γενικά να παραπέμψουμε στην ομολογία του δικαστηρίου. Πρέπει να γνωρίζετε κύριοι βουλευτές ότι υπάρχει μία περίπτωση, η περίπτωση Σοϊσάλ όπου πρέπει να εφαρμόσουμε την απόφαση και του χρόνου θα υπάρξει και υπόθεση Ντεμιρκάν. Με σύμφωνη γνώμη λοιπόν του Κοινοβουλίου, εμείς θέλουμε να γίνει παραπομπή εδώ στην ομολογία του δικαστηρίου. Ένα από τα πιο δύσκολα και αμφιλεγόμενα θέματα που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή είναι η ρήτρα της διασφάλισης. Εμείς θα θέλαμε να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα προσωρινής επαναφοράς. Μερικές χώρες μέλη μπορεί να προσφύγουν στην Κομισιόν και να πούν ότι έχουν συγκεκριμένα προβλήματα ας πούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα γίνεται οτιδήποτε αυτόματα. Η Κομισιόν θα κρίνει την κατάσταση κάθε φορά ανα περίπτωση. Οι θεωρήσεις δεν πρέπει να θεωρηθούν σαν ένα από τα εργαλεία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, ούτε εφαρμογής της πολιτικής του ασύλου. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα της θεώρησης σχετίζεται και με το θέμα του ασύλου και με το θέμα πιθανών κινδύνων προς τη δημόσια ασφάλεια. Γενικά όμως οι σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες για τις οποίες συζητάμε και η συνεργασία στα πλαίσια του Frontex και της Europol είναι θέματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να λύσουμε το πρόβλημα γενικά δεν έχουμε την πρόθεση να ξεπεράσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Σε μεγάλο βαθμό λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το κείμενό της απλώς θα διορθωθεί και δεν θα ξεπεράσουμε τις προτάσεις της. Για την επιτροπολογία από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχουν και πολλαπλές δυνατότητες. Απλώς η προσωρινή επαναφορά του καθεστώτος των θεωρήσεων θα λυθεί με συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά επαναλαμβάνω, τίποτε δεν προτείνεται που να μειώνει τις δικαιοδοσίες του. Ούτε και από την προσθήκη 1 και 2. Με συγχωρείτε που μίλησα πολύ, ήθελα να σας πληροφορήσω πλήρως. Ναι, ευχαριστούμε κύριε Γεζίνσκι. Τώρα η Κομισιόν μήπως θέλει να προσθέσει τίποτα. Όχι, ε, τότε εσείς πάλι κύριε μέρα. Αν θέλετε να συνεχίσετε με την παρέμβασή σας, να ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον κύριο Γιασίνσκι, τον πρόσωπο του Συμβουλίου, για τα τελευταία του σχόλια. Συνεχίζουν να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που είχαμε ήδη κατά νου δεν ε, πρόκειται ακριβώς για τις τεχνικές ε, πτυχές που προκύπτουν από την εφαρμογή της ε, ρήτρας διασφάλισης, αλλά υπάρχουν δύο θέματα που είναι αργώς είναι το θέμα της αμοιβαιότητας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εγκύτητες, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα κράτη-μέλη ή κάποιο συγκεκριμένο κράτος μέλος που δεν το αναφέρω, δεν έχει επιληθεί το θέμα αυτό. και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η στήριξη σε ποσοτικά επίπεδα που θα μπορούσε να έχει αυτή η απόκληση του συγκεκριμένου κράτους μέλους και δεν θέλω να το κατανομάσω. Και νομίζω ότι περιμένουμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα της Τουρκίας, περιμένοντας ε, την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εμένα με ανησυχούν τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από τα ποσοστά που θα εφαρμόζονται σχετικά με τη ρήτρα διασφάλισης. Γιατί δεν είναι μια ανησυχία που είναι μόνο δική μου, αλλά και της κυρίας Λάσπορτ, που δεν τη βλέπω εδώ. Αλλά υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που επίσης ημερίζονται την ανησυχία αυτή όταν καθορίζουν ποσοστά. Έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να ακούσουμε ή να ξανακούσουμε το Συμβούλιο και την Κομισιόν τι πιστεύουν σε σχέση με τα ποσοστά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην ενδεχόμενη εφαρμογή της ε, ρήτρα διασφάλισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Τάνια Φαγιόν, καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και την Πολωνική Προεδρία. Καταρχάς θα ήθελα να δεχτώ την πρόθεση που εκδήλωσε η Κομισιόν για τη ρήτρα ασφαλείας. Την προσωρινή δηλαδή επαναφορά του καθεστώτος των θεωρήσεων. Μόνο όμως σε εξαιρετικές και επίγουσες περιπτώσεις και με δικαιολογημένη αίτηση. Τα κράτη-μέλη έχουν εκφράσει ορισμένες αντιρρήσεις και έχω και ίδια κάποιες αμφιβολίες. Όπως έχει η πρόταση τώρα, το Κοινοβούλιο θα έχει μόνο επεξηγηματικό ρόλο. Το Συμβούλιο, οι χώρες μέλη, δεν χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους την γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου και αυτό είναι αράδεκτο διότι με το Συμβούλιο και την Κομισιόν έχουμε συμφωνήσει ότι πρόκειται για συναπόφαση ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τροποποίηση του κανονισμού και αυτήν τη δικαιοδοσία μας δεν μπορούμε να την εγκαταλείψουμε ούτε μπορούμε να αφήσουμε τις χώρες μέλη από μόνες τους να αποφασίζουν πότε θα επαναφέρουν και πότε όχι το σύστημα των θεωρήσεων. Γιατί έτσι μια χώρα μέλος θα μπορούσε να αρχίσει μια διαδικασία κατάργησης ή άρσης του, του καθεστώτος των θεωρήσεων ε, εφόσον βέβαια υπάρχουν ορισμένοι όροι τουλάχιστον 50% αύξηση σε 6 μήνες παρανόμης μετανάστευσης ή ετοιμάτων ασύλου κλπ. Αυτά λέει η πρόταση. Αλλά αυτό το 50% που λέει είναι πολύ αμφισβητήσιμο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ ψηλό ή πολύ χαμηλό ποσοστό. Από τα στοιχεία που έχουμε από πέρσι και φέτος μπορεί η Γερμανία ανα πάσα στιγμή να επικαλεστεί αυτή την κατεπίγουσα διαδικασία. Γι' αυτό αυτό το 50% είναι αμφισβητήσιμο και χρειάζεται περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την Κομισιόν, μπορεί εκείνοι και τα κράτη-μέλη να παγώσουν το σύστημα των θεωρήσεων χωρίς γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους στην Επιτροπή μας να ζητήσουν να παίξει περισσότερο ρόλο το Κοινοβούλιο. Ελπίζω η ρήτρα αυτή να μην χρειαστεί ποτέ, είναι πολιτικό το θέμα και όπως μας είπε και η Πολωνική Προεδρία είναι τελείως έκτακτο μέτρο που δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε πολύ λεπτά προβλήματα. Τα τέλη του 2009 είχε καταργηθεί το σύστημα των θεωρήσεων για τρεις χώρες των Βαλκανίων και ο αριθμός των αιτητών ασύλου αυξήθηκε και ακόμα και φέτος υπάρχουν τέτοιες αυξήσεις από τη Σερβία και τη Μακεδονία λέει ο Μιλήτρια. Αλλά αφού προσωρινά ζητιούνται τέτοιες εξαιρέσεις, οι λαϊκιστές εκμεταλλεύτηκαν τα πράγματα και άρχισαν τα κράτη-μέλη να περιορίζουν την ελευθερία διακίνησης στο χώρο του Σέγγεν. Εμείς θέλουμε η κατάργηση των θεωρήσεων να είναι μια χειρονομία καλής θέλησης για να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική συνεργασία. Όχι, δεν είναι σκοπός μας να δυσκολέψουμε τα πράγματα για τις χώρες που ήδη είχαν υποφεληθεί από αυτό το σύστημα και τώρα το ξανακαταργούν. Ευχαριστούμε η κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τον εισηγητή Διασδεμέρα και τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας για τις αποσαφηνήσεις τους. Η ομάδα μας υποστηρίζει γενικά την πρόταση, τη θεωρία αναγκαία την εξαίρεση, αλλά ο μηχανισμός που προβλέπεται δεν είναι ίσως ο καλύτερος και πρέπει να ξανασυζητηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα επιβάλλεται η άρση της κατάργησης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν οι προτάσεις αυτές είναι σωστά τεκμηριωμένες. Ιδιαίτερα αυτό το ποσοστό του 50% γιατί τα ποσοστά ποτέ δεν δίνουν ακριβείς αριθμούς προσώπων. Μπορεί να αφορά δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπων. Και αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα. Ανάλογα με το αν μιλάμε με ποσοστά ή απόλυτους αριθμούς ανθρώπων που παράνομα διαμένουν σε ορισμένες χώρες και μέλη. Εκτιμώ λοιπόν το γεγονός ότι το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να δεχτεί το ρόλο που πρέπει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να υπάρξει καλύτερη και περισσότερη συνεργασία για το θέμα μεταξύ μας. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ αναφέρομαι σε μία ρήτρα η οποία θα μπορέσει σε ειδικές περιπτώσεις να διακόψει τη χορήγηση βίζας σε ειδικέ περιπτώσεις. Θεωρώ ότι είναι αυτό ένα καλό μέτρο και μια ε, τέτοια πρόταση θα έπρεπε να έχει ε, ισχύσει και για τις τρίτες χώρες που δεν σέβονται την ε, αρχή της αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη είναι αποτελεσματική και ε, ε, αποτελεσματική και έχουμε λίγες περιπτώσεις μη συμμορφώσεως ε, αλλά σας υπενθυμίζω ότι πέραν των 100 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποφέρουν από την μη εφαρμογή της αλληλεγγύης και η μελέτη της Επιτροπής το είδε και σήμερα. Η τάση αυτή να θεωρούμε την κατάσταση λιγότερο σοβαρή από ό,τι είναι δεν είναι αποδεκτή και θα έπρεπε με τις δύο αυτές χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι πιο αποδοτική στις συζητήσεις της ιδίως όσον αφορά την πολιτική των θεωρήσεων διότι χρειαζόμαστε ένα μέτρο το οποίο θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντίπεινα σε περίπτωση που δεν ισχύσει η ελληνική και να βασιζόμαστε σε αντικειμενικά στοιχεία διότι ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά και είδαμε προσφάτως σε σημαντικές αποφάσεις ότι δεν υπήρξε η σωστή αντίδραση. Η κυρία Ρόιτοβα. Ευχαριστώ. Um, uh, Δεν υπήρξε μετάφραση, κυρία Ροϊτοβά. Μπορείτε να ξαναρχίσετε, παρακαλώ, γιατί είχαμε κάποιο προβληματάκι. Λοιπόν, συμφωνώ με όλα αυτά τα οποία ελέγχθησαν και επίσης με τις επιπλήξεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και προς ορισμένα κράτη-μέλη. Θέλω όμως κάτι να προσθέσω ότι 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών ε, υπόκεινται στην υποχρέωση της θεώρησης παρόλο που ε, οι πολίτες των αντιστοίχων χωρών έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση αναφέρουμε στην Τσεχία. Στην αρχή ε, πριν την ε, προσχώρησή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειαζόμασταν θεώρηση αλλά εδώ και τόσο καιρό δεν κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τον Καναδά. Θα έπρεπε να μας εκπροσωπήσει και να εξασκήσει τις εξουσίες και να εφαρμόσει τις αρχές που θα ίσχυαν αν δεν συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το πρόβλημα είναι σαφώς πολιτικό και πολύ σωστά είπε ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρχει μία ε, ρήτρα διαφυγής αν ε, μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να διατυπώσω μία πρόταση στα κράτη-μέλη. Δηλαδή όταν ένα κράτος μέλος ε, υφίσταται ε, την υποχρέωση θεώρησης μονομερός θα πρέπει να υπάρξει μία περίοδος τριών μηνών προτού αποφασίσει να προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα πρέπει να έχει μία σαφή ημερομηνία ως τελική προθεσμία τρεις-τέσσερις μήνες για να αναλάβει δράση. Βεβαίως θα μπορεί να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ε, να ανατραπεί η θέση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε 27 μήνες όπως στην περίπτωσή μας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει αποδεχθεί πλέον του ενός έτους τώρα την θέση της χώρας μου και δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση. Ε, ναι μεν ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λύσει τα προβλήματα αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε εμπιστοσύνη διότι το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης σε μία αρχή η οποία να βασίζεται στην ελληνική και παρακαλώ να με στηρίξετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την Τουρκία ουσιαστικά. Διότι την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο η ε, Επίτροπος μάλιστα μας έκανε ε, μία αναφορά σχετικά με τις θεωρήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι προτίθεστε να κάνετε στο θέμα αυτό ε, και πέραν αυτού. Εδώ και δύο χρόνια Έχουμε σκεφτεί να κάνουμε ε, μία έρευνα και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με την ε, υποχρέωση θεωρήσεων και να ανατρέξουμε στο 1972, δηλαδή ποιες χώρες τότε είχαν υποχρέωση θεώρησης. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, βλέπω ότι τώρα έχει επανέλθει ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αίθουσα. Μπορώ να δώσω το λόγο ε, στον εκπρόσωπο πρωτού, ε, δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλους παρακαλώ εξηγήστε μου γιατί έχουμε αυτό το, αυτά τα ποσοστά στην πρόταση που διατυπώσαμε. Καταρχήν σας προτείνουμε την αρχή της επιτροπολογίας και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε οριοθετημένα κριτήρια κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να ε, ε, ισχύσει η ε, ρήτρα διαφυγής η οποία θα είναι το τελευταίο μας καταφύγιο για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε των περιστάσεων. Χρειαζόμαστε αυτά τα ποσοστά διότι όντως όπως σας λέω πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί η ε, διαδικασία επιτροπολογίας που επιτρέπει μία γρήγορη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι στην τρίτη παράγραφο της προτάσεως για τη ρήτρα διαφυγής λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει την κοινοποίηση του κράτους μέλους, θα σταθμίσει πόσα κράτη-μέλη επηρεάζουν από, αυτήν, την, από αυτό το μέτρο και ε, θα εξετάσει την κατάσταση της, ε, των μετακινήσεων εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο νικητούμε κοιτάμε και τις επιπτώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο σημαίνει, για να αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι αν έχετε σε ένα πολύ μικρό κράτο, κράτος μέλος μόνο τρία άτομα τα οποία ζητούν άσυλο, το οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα γίνουν έξι, έχετε μια αύξηση 100%. Αλλά ε, θα κοιτάξουμε τις συνθήκες και θα πούμε, αλλά εδώ μιλάμε μόνο για ένα κράτος το οποίο έχει μία αύξηση 100%. Άρα καλύπτει τα κριτήρια, τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια, αλλά αυτό δεν επαρκεί για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την ρήτρα διαφυγής διότι ε, πρόκειται ε, παραδείγματος χάρη μόνο για ένα κράτος το οποίο έχει ελάχιστους ετώντες άσυλο. Γι' αυτό και πάντοτε θέλουμε να εξετάσουμε τη συνολική ε, επίπτωση αυτών των συνθήκων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την Τουρκία. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξή μας, αλλά ε, επιτρέψτε μου να πω τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή ότι θα προσπαθήσουμε να, κάνουμε, ε, να προσφέρουμε διευκολύνσεις θεωρήσεων στους Τούρκους πολίτες ε, στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και ε, του κώδικα θεωρήσεων που μας δίνει κάποια ευελιξία για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις να αυξήσουμε ε, τον αριθμό των θεωρήσεων ή να εξετάσουμε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Αυτό εννοούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μίλησε για διευκολύνσεις, δηλαδή δεν πρόκειται για για την ε, συμφωνία διευκολύνσεως των θεωρήσεων που έχουμε ε, ε, με ορισμένες χώρες οι οποίες είναι στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, είναι σαφές τι εννοούσαμε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ουσιαστικά δύο χώρες ε, ε, μπλέκονται ε, στο θέμα αυτό, οι άλλες δεν πλήττονται και γι' αυτό εάν κοιτάξετε την πρότασή μας για την ε, ε, τροποποίηση του 539 θα δείτε ότι προσπαθούμε να αναμορφώσουμε ε, τις κοινωνικές διατάξεις στην απόφασή μας για την Τουρκία και αυτή τη στιγμή θα ήθελα να περιοριστώ εδώ αλλά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω και σε άλλα ερωτήματα εάν μου τεθούν. Ο κύριος Δίας Διονέρα τώρα για να κλείσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ε, κυρία Φαγιάννα Καλένσιου, κυρία Ρεϊτόβα και την κυρία Μποσκούρ για τις παρεμβάσεις τους. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε και ένα ανησυχίε. Αφενός ε, λέγεται ότι για να αποφύγουμε καταχρήσεις και να διευκολύνουμε την ε, κυκλοφορία των νόμιμων μεταναστών ε, θα χρειαζόταν η εφαρμογή αυτής της ρήτρας διασφάλισης. Όμως υπάρχουν ε, κάποια θέματα και τεχνικά αλλά και πολιτικού χαρακτήρα. Για να συνοψίσω, τα θέματα που έχουν πολιτικές αποκρόσεις έχουν περισσότερο να κάνουν με την εφαρμογή του θέματος της αμοιβαιότητας και ε, το θέμα της αμοιβαιότητας, ε, όπως μας είπε η κυρία Ρουιτόβα, θίγει κυρίως την τσεχική δημοκρατία και τις σχέσεις της με τον Καναδά. Και αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει επιληθεί, είναι επιτάπητος και είναι ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης να σκύψουμε και θα πρέπει να το συζητήσουμε και με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν, καθώς ακόμη δεν έχει ανοίξει προθεσμία για την παρουσίαση τροπολογιών, για την κατάσταση τροπολογιών, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε αυτό το θέμα για να προσπαθήσουμε να ξεβρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα, στο οποίο αναφέρθηκαν όλοι οι συνάδελφοι, που πήραν το λόγο, έχει να κάνει με την εφαρμογή των ποσοστών τη στιγμή της χρήσης ε, της ρήτρας ε, διασφάλισης. Μπορεί όταν εκπονούμε την έκθεση ίσως να μπορούσαμε να μιλάμε για νούμερα και όχι για ποσοστά γιατί μπορούμε να εμπιστευτούμε περισσότερο τα νούμερα παρά τα ποσοστά. Γιατί αν ε, μιλάμε το χάρη ε, ε, 4 8 άτομα θα, θα είχαμε 100%. Αν μιλάμε όμως για 4 ή 8 άτομα, είναι κάτι άσχετο. Έτσι λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για ακριβή νούμερα ή κατά προσέγγιση νούμερα, παρά για ποσοστά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε και κατόπιν να το θέσουμε στη συζήτηση με το Συμβούλιο και το Κομισιόν. Και σε σχέση με την παρέμβαση της Κομισιόν, ναι, νομίζω ότι είναι σαφής η διαδικασία. Είναι σαφές πως ε, όταν ε, έχουμε κοινοποίηση από ένα κρατός μέλος, τότε θα πρέπει να αξιολογηθούν ε, κάποιε συγκεκριμένε συνθήκη, λαμβάνοντα υπόψη διάφορε εκθέσει, μεταξύ των οποίων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και η έκθεση της Frontex και η έκθεση του ΕΑΣΟ. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που υπόκειται σε σχέση με τα, ε, υπάρχει σε σχέση με τα άλλα δύο. Ο ρόλος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπολογία, είναι ένα θέμα κατανοητό για να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες ε, ανάγκες, τις έκτακτες περιπτώσεις. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρχει και ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα σε όλα αυτά. Ο κ. Στακούστη μας είπε ήδη ότι υπάρχει δέσμευση να είναι σε μόνιμη επαφή με το Κοινοβούλιο κάθε φορά που κατά εξαίρεση θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αυτή η ρήτρα διασφάλισης. Όμως ε, σε αυτή την έκθεση θα μπορούσαμε κι εμείς ε, να αναγράφουμε αυτή τη διάθεση της Κομισιόν. Θα μπω στο χειρουργείο την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Δευτέρα θα χειρουργηθώ. Έτσι λοιπόν δεν θα είμαι διαθέσιμος για μια εβδομάδα, όμως στις 20 του μήνα ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με την αξιολόγηση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστούμε κυρία Δίας Δαμέρα για την παρουσίαση και για τα καταληκτικά σας σχόλια και σας εύχομαι ε, περαστικά να πάει πολύ καλά το χειρουργείο σας, δεν το γνωρίζαμε και να επανέλθετε εδώ πολύ σύντομα για τις εργασίες μας ε, στην Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ό,τι καταλαβαίνω θα παρουσιάσετε την έκθεσή σας, το σχέδιο έκθεσης στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Λίμπες τον Νοέμβριο. Ωραία μάλιστα. Λοιπόν, καλούνται και οι σκιώδεις. Ε, κύριε Συγγνώμη που παρεμβαίνω αμέσω μετά τον εισηγητή, αλλά θέλω να κάνω μια μικρή διευκρίνηση σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, ιδιότητας. Δεν είναι μόνο ε, η Τσεχική Δημοκρατία που έχει αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε για 15 κράτη-μέλη. Πολωνία, Βουλγαρία, Κύπρος, 5 μέλη, 5 κράτη-μέλη δεν επωφελούνται. Μάλιστα. Ο κ. Διασδομέρη για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ τον κύριο Έντσιου για τη διευκρίνηση αυτή. Να σας πω ότι γνωρίζω όσα λέτε. Απλώς ε, Αναφέρθηκα στην Τσεχική Δημοκρατία μόνο και στο πρόβλημα που έχει με τον Καναδά. Επειδή το έθιξε η κυρία Ρόιτοβα. Αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλα κράτη-μέλη μεταξύ αυτών και η Ρουμανία. Η χώρα του συναδελφού που ζήτησε το λόγο πριν. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε Δία Θα τα ξαναπούμε λοιπόν εδώ. Ας περάσουμε στο σημείο 10 που είναι το σημείο 3 στην ε, ε, ημερήσια διάταξη, είναι θεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Έχουμε την κυρία Φλότρο ως εισηγήτρια. Εξετάζουμε τις τροπολογίες και τι φαίνεται τώρα Η ημερομηνία για την κατάσταση των πολυγόνων ήταν η 14η Σεπτεμβρίου και τώρα βρισκόμαστε εδώ ακριβώ για να συζητήσουμε τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Και θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στην κύριο Φλότρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχήν τους συναδέλφους γιατί κατατέθηκαν 71 τροπολογίες σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότης από όλες τις πολιτικές ομάδες. Τους ευχαριστώ γιατί οι περισσότερες από αυτές τις τροπολογίες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την θέλησή μας να ανανεωθεί η πολιτική γειτονία, ιδίως ως προς την κυκλοφορία των προσώπων, τη μετανάστευση και τον έλεγχο αυτής. Πολλές τροπολογίες τις δέχομαι, αλλά αφορούν μάλλον την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας όπως θα τη συζητούσε η Επιτροπή Εξωτερικών από άποψη εξωτερικών. Για μας χρησιμότερο θα ήταν νομίζω να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στο δικό μας θέμα ανθρώπινα δικαιώματα, άσυλο, μετανάστευση και γι' αυτό ίσως αντιταχθώ σε ορισμένες τροπολογίες χωρίς να είμαι αντίθετη με το πνεύμα τους. Επίσης είμαι ικανοποιημένη γιατί για τους περισσότερους συναδέλφους η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων είναι κάτι που το δέχονται γιατί αν το ανταποκρίνεται στο θέμα, στο πρόβλημα της κινητικότητας και των νέων δικαιωμάτων όπως προκύπτουν από τα τελευταία γεγονότα στο νότο της Μεσογείου. Για την παράγραφο 4 σημείωσα ότι ορισμένοι συνάδελφοι ήθελαν και συμφωνώ και εγώ να προσθέσουμε παραπομπή και σε άλλες συμβάσεις συμφωνίες όπως το πρωτόκολλο για, για το δουλεμπόριο δεσμευτικά κείμενα και μέτρα δηλαδή για τη συμφωνία για τα δικαιώματα των μεταναστών και των οικογενειών τους είναι κάτι σημαντικό γιατί η συμφωνία αυτή, η σύμβαση αυτή δεν προβλέπει καινούργιες υποχρεώσεις για τα κράτη-μέλη αναφέρει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις των μεταναστών και μεταναστριών και την έχουν ήδη δεχτεί πολλές χώρες από το νότιο τμήμα της Μεσογείου. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει και τα κράτη της Ένωσης καθεαυτά να την εγκρίνουν, να την επικυρώσουν. Μου φαίνεται κάτι λογικό και σημαντικό αφόσον μάλιστα βρισκόμαστε σε περίοδο συζήτησης με τις χώρες αυτές που είναι στο δρόμο του εκδημοκρατισμού. Η παράγραφο 5 για τα ευρωπαϊκά ταμεία εδώ, Γι' αυτά υποστηρίζω ότι τροπολογία ζητάει καλύτερα στοχευμένη χρήση των ταμείων. Περίπου όπως ανακοινώθηκε και την περασμένη εβδομάδα από την Κέτι Άστον μετά την επίσκεψή της στην Τουνησία που ζήτησε το ξεπάγωμα 4 δισεκατομμυρίων. Είναι πολύ σημαντικό και οι κοινοβουλευτικοί να απαιτήσουν να υπάρχει έλεγχος της δαπάνησης αυτών των ποσών για την στήριξη του εκδημοκρατισμού και της οικονομικής ανάπτυξης ε, αλλά και της κοινωνικής ισότητας όπως ακριβώς ζητούσαν οι εξεγερμένοι. Υπάρχει επίση ένα θέμα με, για την εταιρική σχέση με, την κοινωνία, με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και εδώ συμφωνούμε. Η νέα πολιτική γειτονία θα έχει και νέα ποιοτικά κριτήρια μεγαλύτερος ρόλος θα υπάρχει δηλαδή από τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ μπορούμε να ζητήσουμε να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα γίνει κάτι τέτοιο ως προς την επιτήρηση της εφαρμογής, συζητήσεις, συνεννοήσεις κλπ. Αυτό που θέλουμε πάντως είναι η κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει περισσότερο σε όλα τα επίπεδα της εφαρμογής της αναθεωρημένης πολιτικής γειτονίας. Τέλος υπάρχει και η παράγραφος για την κρίση των προσφύγων όπως συζητήθηκε και από την Ολομέλεια και εδώ νομίζω ότι εδώ μπορούμε να βρούμε επίσης πολύ ευρεία συνένεση για να υποστηρίξουμε συγκεκριμένα μέτρα όπως να ζητήσουμε οι έρευνες για τα ανθρώπινα δράματα που σημειώνονται να τελειώσουν επιτέλους και να μας δηλώσουν αν η Ιταλία έχει καταλήξει πλέον τις συνεννοήσεις της με τη Λιβύη και την Τινησία να γίνουν δημόσια όλα αυτά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τις πόρτες της στους αιτητές ασύλου και τους πρόσφυγες που έχουν μπλοκαριστεί, που είναι μπλοκαρισμένοι αυτή τη στιγμή ακόμα στη Λιβύη, αλλά και στην Τινησία και την Αίγυπτο, πρέπει το πρόγραμμα επανεγκατάστασής τους να εφαρμοστεί. Αυτή είναι η παράγραφος που αφορά περισσότερο την σημερινή συγκυρία και επικαιρότητα. Και εδώ νομίζω δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που δέχομαι και μπορώ να τις δεχτώ ως έχουν, δεν είναι τροποποιήσεις των υπαρχουσών παραγράφων, αλλά νέες παράγραφοι. Δεν θέλουμε βέβαια να γίνει πολύ μακροσκελής και χαόδη ε, χαόδης η γνωμοδότησή μας, ούτε να επικαλυφθεί με τα θέματα της ΕΠΕΞ. Αύριο στις 11 θα το συζητήσουν εκείνοι και μετά από τη συζήτηση θα γίνει τώρα. Θα ήθελα σήμερα το απόγευμα να προτείνω συμβιβασμούς για να προχωρήσει το πράγμα και να είμαστε έτοιμοι για αύριο. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη συζήτηση σχετικά με τις τροπολογίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν η κυρία Νεντέλτζεβα. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια ε, και για τις τροπολογίες διότι είναι τροπολογίες με τις οποίες συμφωνούμε επί της ουσίας αλλά νομίζουμε ότι δυσχεραίνουν το κείμενο και πρέπει αυτή η γνωμοδότηση να είναι όσο δυνατόν ο πιο ευέλικτη γι' αυτό και συμφωνώ να υπάρξουν συμβιβασίες τροπολογίες και έρχομαι στο δεύτερο σημείο που συμφωνώ ε, με την εισηγήτρια να παραμείνουμε στην Επιτροπή μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή τους ε, αύριο θα υπάρξει μία συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και εν ονόματι του ΕΛΚ έχουμε διατυπώσει ορισμένες προτάσεις που θα θέλαμε να αντικατοπτρίζονται στη συμβιβαστική λύση, δηλαδή κινητικότητα των ε, μεταναστών, δεύτερον ε, το, την αντιμετώπιση του κινδύνου της ε, διαφυγής των εγκεφάλων των εξύπνων και μορφωμένων προς άλλες χώρες, επίσης καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας και ένα τέταρτο θέμα είναι να ε, κάνουμε ε, ε, μία επανεφαρμογή της κινητικότητος για τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς. Ε, θα πρέπει να υπάρχει επίσης ένας ανθρωπιστικός ε, διάδρομος που θα πρέπει να καταρτιστεί προς την Τουρκία, ε, τη Λιβύη και την Συρία και έχω και ακόμη δύο σημεία για τα οποία επιφυλάσσομαι εν ονόματι του ΕΛ και σχετικά με την τροπολογία 16 για την ενισχυμένη συνεργασία στις συμφωνίες επανεισδοχής και και ε, το μορατόριο στις ε, συμφωνίες ε, επανεισχωρήσεως. Κατά τα άλλα είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις και όπως είπα συμφωνώ με την εισηγήτρια για να καταλήξουμε σε μία γνωμοδότηση η οποία θα αναβιώσει την πολιτική γυτνιάσεως την οποία χρειαζόμαστε αλλά πρέπει πρέπει να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τις δυνατότητες επιτυχίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα διότι η πολιτική γυτνιάσεως είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται πάρα πολύ μετά τα γεγονότα στη Βόρειο Αφρική. Χαιρετίζω λοιπόν την ε, έκθεση της Επιτροπής ΑΦΚΟ και τη δυνατότητα να ε, καταρτήσουμε μία γνωμοδότηση την οποία συνέταξε η κυρία Φλότερ. Πιστεύω όμως ότι είναι σημαντικό αυτή η Επιτροπή να μπορέσει να καλύψει την εντολή της και να επικεντρωθεί στις αρμοδιότητές μας αντί να κάνει μια πολύ ευρία γνωμοδότηση πιο ενδιαφέρουσα ίσως αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε περισσότερο και γι' αυτό πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα για το τι μας απασχολεί. Οι ορισμένες τροπολογίες είναι πολύ ασαφές, ασαφείς και αναφέρονται σε άλλα θέματα τα οποία χρειάζονται περισσότερο χώρο και περισσότερη εμβάθυνση για να μπορέσουν να αποδώσουν θα πρέπει να ε, στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή ΑΦΚΟ σχετικά ε, με τις αρμοδιότητές μας επί ε, των μετακινήσεων του ασύλου και τις επανατοποθετήσεως διότι προσπαθούμε να έχουμε μία συνεκτική και σύντομη γνωμοδότηση και να αποφύγουμε να πλατιάσουμε. Ε, αύριο θα συμμετάσχω στην ε, συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε επιτυχίες συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ. είμαι πολύ σύντομος ε, στην παρέμβασή μου. Εγώ συμφωνώ με όσα είπαν οι συνάδελφοι, κυρίως οι τρέκοι συνάδελφοι ε, Wilson και τα λοιπά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι για να μπορέσουμε να δώσουμε ξεκάθαρα μήνυματα για, από την προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων μέχρι και τα δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά και υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούνται και από τους ε, μετανάστες ε, και πρέπει να υπάρχει κοινωνική ισότητα. Έχω κάποια αμφιβολία σε σχέση με το αν οι θεωρήσεις ε, στο στάδιο αυτό μπορούν να αποτελούν ένα χρήσιμο στοιχείο σκέψης, προβληματισμού, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό να λαμβάνουμε υπόψη και τα ευρωπαϊκά και κονδύλια που χορηγούνται για την αξιολόγηση αυτών των σχέση συνεργασίας. Ο στόχος βέβαια πρέπει να είναι σαφής η Ευρώπη. Θα πρέπει να δείχνει αλληλεγγύη στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Έτσι λοιπόν οι συμφωνίες θα πρέπει να συνάπτονται απευθείας από το ευρωπαϊκά όργανα, διμερείς ε, συμφωνίες ε, και εμπορικές ε, συμφωνίες στο πλαίσιο των συμφωνιών πλαίσιων καθορίζουν ποια είναι και τα καθήκοντα και υποχρεώσει των τρίτων χωρών ε, και στο πλαίσιο της απαραίτητης ε, αστυνομικής συνεργασίας προκειμένου να ε, έρχονται στην Ευρώπη όσοι πραγματικά έχουν δικαίωμα. Δηλαδή να έχουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και προσφύγων. Επίσης πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, των συμφωνιών επανεισδοχής. Εμείς ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά και φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γρούτσας. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ την κυρία Φλότρ ε, για τη δουλειά της και όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Και καθώς αύριο θα έχουμε τη συνεδρίαση των ε, σκεδών συγγητών, θα κάνω μόνο μια γενική παρατήρηση. Όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρισκόμαστε σε μια δύσκολη και ευαίσθητη κατάσταση, λεπτή κατάσταση, γιατί αφενός ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ευρωπαίους πολίτες αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση, την, ε, η ανασφάλεια που έρχεται από αυτή την οικονομική κρίση και φυσικά φαινόμενα όπως αύξηση της ξενοφοβίας εμφανίζονται και πάλι και φυσικά ε, ορισμένοι το εκμεταλλεύονται πολιτικά αυτό. Από την άλλη βλέπουμε σημαντικές αλλαγές ε, στην γειτονιά μας, στη Βαλκάνια, στην Κεντρική Ασία, στο ο και κυρίως στην Βορειοαφρική, στον Αραβικό κόσμο. Αυτό δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευκαιρία να διαδραματίσει ένα ρόλο, να έχει αυξημένο ρόλο και να επηρεάσει την ε, δική της περιοχή και τολμώ να πω ότι πρέπει να δούμε τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της ως επένδυση για το μέλλον. Παραδείγματο χάρη, το να έχουμε μια καλή μεταναστευτική πολιτική σήμερα σημαίνει ότι θα αποφύγουμε τεράστια προβλήματα για την Ευρώπη στο αγγί μέλλον. Ποιο αμφιβάλλει ότι η Ευρώπη θα ε, αντιμετωπίσει μαζικέ μεταναστευτικέ ροέ που δεν θα μπορούν να, να ελεγχθούν στο μέλλον αν δεν αναλάβουμε τώρα την απαραίτητη δράση και προέρχομαι από την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε έχουμε πολύ συγκεκριμένη εμπειρία με το θέμα αυτό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να διατηρηθούν ευαίσθητες ισορροπίες στο θέμα αυτό, γιατί οι Ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς και απειλούνται είναι ευάλωτη απέναντι σε λαϊκιστικές προσεγγίσεις, κυρίως ως προς τα θέματα αυτά. Έτσι λοιπόν, ε, θα ήθελα να έχουμε μια καλή συνεργασία με τις άλλες ομάδες και θα ξεκινήσουμε αύριο αυτή την καλή συνεργασία με τη συνάντηση των σκανδών Μάλιστα, ευχαριστώ κύριο Τριανταφυλλίδης. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συμφωνώ και εγώ με άλλους συναδέλφους για τη σημασία που έχουν προσδώσει σε αυτή την έκθεση ιδιαίτερα μέσα στις ε, συνθήκες τις σημερινές όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την Αραβική Άνοιξη. Είναι γι' αυτό που και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, την κυρία Φλότ, για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε εντός ομολογουμένως πολύ περιορισμένων συνθήκων, διότι το να κατορθώσει ένας να αναφέρει όλους τους σημαντικότερους στόχους που θα έπρεπε να έχει η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας σε μια και μόνο σελίδα είναι μια μεγάλη πρόκληση μέσω των τροπολογιών μας σε ό,τι αφορά το δικό μας και δική μας την ομάδα προσπαθήσαμε να στηρίξουμε την προσέγγιση της ε, εισηγήτριας προσθέτοντας ορισμένα στοιχεία που μας φαίνονται κρίσιμα. Και πιο συγκεκριμένα, εάν και η Επιτροπή υποστηρίζει ότι έχει υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση στην πολιτική γειτονίας που βασίζεται σε μια πιο ίση εταιρική σχέση με σαφείς όρους, Εν τούτης θεωρούμε σημαντικό να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι οι νέες προτάσεις της Επιτροπής συνεχίζουν να βασίζονται σε μια λογική που συνδέει τη συνεργασία και την παροχή βοήθειας στη δέσμευση της γειτονική χώρας να καταπολεμά αποτελεσματικά την παράτυπη μετανάστευση μέσω εντός των άλλων και της σύναυσης συμφωνιών επανεισδοχής που ισχύουν για υπηκόους τρίτων χωρών παρά το γεγονός ότι αυτό αποτελεί συχνά πηγή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά τα περιλαμβάνουμε στις ε, τροπολογίες που έχουμε υποβάλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. And Mr. Thank you. The report... Ευχαριστώ. Η έκθεση εγκρίνει ε, τους αγώνες για τη δημοκρατία ε, στην νότια αυτή της Μεσογείου και φυσικά εγώ συμφωνώ απόλυτα. Επίσης αναφέρεται στο δικαίωμα της κινητικότητας ως ανθρώπινο δικαίωμα. Πρέπει όμως να αναρωτηθώ γιατί μπήκαν σε τόσο κόπο να μπουν σε τέτοιο κίνδυνο για να καταστήσουν δημοκρατικές τις χώρες τους και να μπορούν να ζουν ελεύθερα χώρες κατά αν εμείς ε, ε, υποθέτουμε και σωστά μάλλον ότι το πρώτο δικαίωμα που θέλουν να ασκήσουν είναι τις μετανάστες στην Ευρώπη είτε επίσημα είτε με μέτρα χαλάρωσης των θεωρήσεων είτε ως πρόσφυγες που θα επιζητούν την ειρήνη και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κυρία Φιλότρη, για τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχουν πολλές ε, ε, παρατηρήσεις οι οποίες δεν συγκλίνουν αλλά θα οριοθετήσουν τουλάχιστον τη μορφή και νομίζω ότι θα χρειαστεί να εγκαταλείψουμε ορισμένες τροπολογίες και ορισμένες παραγράφους και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι διότι για μένα είναι βασικό να ε, έχουμε και να παρουσιάσουμε το νέο δικαίωμα στην κινητικότητα το οποίο πρέπει να βασίζεται στις διεθνείς συνθήκες. Μπορεί ο καθένας να εγκαταλείψει τη χώρα του. Αυτό είναι διεθνές δίκαιο, αλλά δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το κείμενο να εκφράζει αυτό που βλέπουμε και αυτό που θέλουμε να ανανεώσουμε στις συμφωνίες και συνεργασίες. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει με τις νέες κυβερνήσεις που οφείλονται σε δημοκρατικές διαδικασίες, να ανανεώσουμε ε, τις ε, συμφωνίες ε, οι οποίες όμως δεν θα μοιάζουν με αυτές που κράτησαν οι νότιο-αμερικανοί επί χρόνια έναντι της Ευρώπης. Θέλουμε να αναπτυχθούν οι χώρες αυτές και να αυξήσουμε τις συναλλαγές μαζί τους. Είναι λοιπόν ένα βαστικό στοιχείο το οποίο δεν θα ξεχάσουμε ε, ε, αύριο στην ε, συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και θα προτείνω συμβιβαστικές λύσεις για να βασίσουμε εκεί τη συζήτησή μας και ορμόμενη από τη συζήτηση την οποία κάναμε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ κυρία Φλότρ. Και τώρα νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι η η ψηφοφορία επί του θέματος θα γίνει 17 ε, Οκτωβρίου και ε, αυτό μας φέρνει στο τελευταίο σημείο μετά από την ώρα της ηλεκτρής ε, ψηφοφορίας. Προβλέπεται όμως ε, στις 11 η ώρα να ξεκινήσει η ψηφοφορία και επειδή πολλά, ε, ε, πολλοί ευρωβουλευτές έχουν κανονίσει τα ραντεβού τους μέχρι τις 11 να κάνουμε μία διακοπή για 10 λεπτά και όσοι δεν έχουν την ηλεκτρονική τους κάρτα μαζί μπορούν εντωμεταξύ να φροντίσουν να την προμηθευτούν που θα χρειαστούμε για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και στη συνέχεια διότι θα έχουμε ψηφοφορίες ε, κοινέ με την Επιτροπή Γυναικών ε, για τα κοινά μας θέματα. Ευχαριστώ.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 Schade, που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 Dear colleagues, if you want to take your seats. Καθίστε παρακαλώ. It's 11 sharp, so we should get... Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε για να μην καθυστερήσουμε κι άλλο. Παρακαλώ να έχετε τις κάρτες σας. Τις έχετε, τις έχετε βάλει στη σχισμή. Ε, τότε είμαστε και έτοιμοι. Το 12, ψηφοφορία, το 13 δηλαδή, της νομοδότησης του κυρίου Μούλιντερ για την κυκλοφορία και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. Για την έγκριση των τροπολογιών μια Κύριε Δία Θεμέρα, έχετε και εσείς την κάρτα σας. Αμέσως τώρα την έβαζα κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω για την κατανόησή σας να μου επιτρέψετε να ψηφίσω ανάταση. χειρός. Μάλιστα, θα προσμετρήσουμε, δηλαδή θα ψηφίσουμε μια ψηφοφορία με ένα τεσχυρός από το ΕΛΚ.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 45 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβασμό 2 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά Αποχέ. εγκρίνεται. 53 υπέρ. Συγγνώμη, ξέχασα νομίζω ότι καταπίπτει. 49. Την ξέχασα. 49 υπέρ. Κατά εποχέ συγκρίνεται. Τώρα. Επιστρέφουμε στην 53 υπέρ. Κατά εποχέ γκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά εποχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 2 δεν έχει καταπέσει. Ψηφίσουμε την υπαριθμόν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 56. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 15 εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 55. Όχι, 57, δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί. 58 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Έχουμε τρία μέρη στην επόμενη υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα αποσύρεται τρίτο τμήμα υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά απορρίπτεται 70 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 71 όχι, έχει καταπέσει 6 και 72 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 7 και 73 ταυτόσιμες υπέρ, κατά εποχές, εγκρίνονται. 8 και 74 υπέρ, κατά εποχές, εγκρίνονται. 76 υπέρ, κατά εποχές, εγκρίνονται. 77 υπέρ, κατά εποχές, απορρίπτονται. Εκτιμώντες, τροπολογία 9 υπέρ, κατά εποχές εγκρίνεται. 10 Επέρ. κατά εποχές εγκρίνεται. Είδα το διπλό ναι. Υπέρ <laughs> εγκρίθηκε. 11 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 15 είδατε. τροπολογία προφορική για το κτιμώντα 7 από τον συγητή υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 16 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται τροπολογία 1 για το κτιμώντα 13 Mm-hmm. Τροπολογία 19. Βλέπω ότι έχει αποσυρθεί το πρώτο τμήμα. Ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κοιτά. Εποχές. Εγκρίνεται. Και 20. Υπέρ. Κοιτά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 47 υπέρ, μία κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Μόλτερ. Thank you. Don't miss the electronic cards because we still be having some... Λοιπόν, θα έχουμε και άλλη ψηφοφορία μεικτή με την Επιτροπή ΦΕΜ για την εντολή προστασίας. Κύριε Κικόδο, έχει το λόγο. Can I please ask you, and you know how scrupulous... Να σας ε, ρωτήσω, Πρόεδρε να ζητήσετε από κάποιον που οργανώνει τα ρολόγια για να τα βάλει στη σωστή αίθουσα. Εγώ ήρθα στην αίθουσα ακριβώς στις 10.59 για την ψηφοφορία ε, των 11. Εσείς είχατε ήδη ξεκινήσει και 5 λεπτά και έδειχνε 11 και 5 το ρολόι, όμως δεν είναι καλό να μην έχουμε συγχρονισμένα ρολόγια. Και εγώ έχασα ορισμένε από αυτές τις ψηφορίες και υπήρχαν και άλλοι που ήρθαν ε, και άλλοι μετά από μένα. Θέλω να συγχρονίσετε τα ρολόγια γιατί εγώ ήρθα εγκαίρος για να ψηφίσω. Α, έχετε δίκιο, δίκιο έχετε. Εγώ έβαλα τα δυνατά μου για να διατηρήσω την ώρα. Μάλιστα έκανα και διάλειμμα 10 λεπτά. Γιατί ολοκληρώσαμε το προηγούμενο σημείο 10 λεπτά νωρίτερα. Και διέκοψα για 10 λεπτά ακριβώ για να ξεκινήσω στις 11 ακριβώς και είδα εκείνο το ρολόι και όταν έδειξε 11 ξεκινήσαμε. Ίσως, δεν ξέρω αυτό το ρολόι, πάει μπροστά, πάει πίσω. Τέλος πάντων θα διασφαλίσω έτσι ώστε να είναι ακριβή τα ρολόγια για να σεβόμαστε όλοι την κατάλληλο ωράριο στις εργασίες της Επιτροπής Λίμπια. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο. Ε? having now, having now a joint debate on the asylum. Τώρα έχουμε κοινή συζήτηση για το πακέτο ασύλου. Και στις 12 Έχουμε 40 λεπτά για αυτή τη συζήτηση και στις 12 θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, με την Επιτροπή ΦΕΜ για την εντολή προστασίας. Και θα έχουμε και άλλη μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αλλά τώρα έχουμε μία συζήτηση για τα σημεία 5 και 13. Για το πακέτο σύλλου. Well, well, well, well. We have another timing issue here. Με και άλλο θέμα εδώ με το χρόνο. Yes, we have another timing issue. The presidency, the Polish presidency. Η Πολωνική Προεδρία θα κάνει μια παρουσίαση. Mm. Ο κύριος ε, Μίλλερ αρχικά επρόκειτο να έρθει, αλλά δεν μπορεί να τα καταφέρει, λυπάται. Και θα έρθει επαρτημών 2 του Υπουργείου, ο Υπουργός. Για θέματα σύλλου ο κύριος Πιότερ Στασάσης. Αλλά μου είπαν ότι έρχεται από το αεροδρόμιο. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν με το χρόνο. I mean, we should get started with his presentation. Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με τη δική του παρουσίαση, έτσι. και μάλλον θα έπρεπε να διακόψουμε για μια ακόμη φορά έτσι ώστε να του δώσουμε την ευκαιρία να φτάσει εδώ. Ας διακόψουμε και πάλι λοιπόν ο Πρόεδρος. Ίσως να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο μας αλλάζοντας στη σειρά των διαφορών στοιχείων της εξίσωσης. Κυρία Γκίον, ως εισηγήτρια θα μπορούσε να πάρει το λόγο. Ίσως να ακούσουμε την κυρία Γκυγιόμ καταρχήν. Και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον ε, Υφυπουργό ε, του Άσυλου. Κυρία Γκυγιόμ, έχετε το λόγο. Oui, merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μου δίδετε τον λόγο για να καλύψω το χρόνο μέχρι του να έρθει ο εκπρόσωπος της ε, Πολωνικής Προεδρίας αλλά καταρχήν εγώ σκεφτόμουν το αντίστροφο διότι νόμιζα ότι ο χρόνος έπρεπε να, γίνει, ε, να διατεθεί σε δύο συζητήσεις καταρχήν ο υφυπουργό να παρουσιάσει την κατάσταση των συζητήσεων και ε, να υπάρχει μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτών των ε, επί αυτών των θεμάτων παρόλο που ο χρόνος ε, είναι πολύ σύντομος. Εγώ θα βοηθήσω λοιπόν παρουσιάζοντας ε, τα στοιχεία της οδηγίας για τη διαδικασία παρόλο που τα στοιχεία φαίνονται ότι είναι σημαντικά και ενδεχομένως θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και να σεβαστούμε το χρόνο που μας έχει διατεθεί και την προθεσμία του 2012. Όταν θα έρθει λοιπόν ο υφυπουργό, θα επανέλθω στο θέμα του ασύλου γενικότερα και στο πακέτο γιατί έχω να κάνω άλλες προτάσεις να κάνω επ' αυτούς και εδώ έρχομαι εις ε, την ε, οδηγία της, ε, τη διαδικαστική η οποία είναι σημαντική για το πακέτο αυτό διότι ίσως θυμάστε ότι παρουσίασε η Επιτροπή μία νέα πρόταση είχαμε την ευκαιρία με τους Σκιώδης να συζητήσουμε με την Επιτροπή επί διαφόρων θεμάτων και όσον αφορά την ουσία θα ήθελα να κάνω ορισμένες αξιολογήσεις και ουσιαστικά να χαιρετήσω την εργασία που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επιτύχει μία ισορροπία μεταξύ των κόκκινων γραμμών που είχε θέσει το Κοινοβούλιο και ε, κάποια ευελιξία σε ορισμένα σημεία προς τα κράτη-μέλη. Η ευελιξία πρέπει να υπάρχει αλλά δεν πρέπει να είναι αντιπαραγωγική διότι πρέπει να επιτύχουμε τον στόχο τον οποίο έχουμε θέσει συλλογικά. Θα επανέλθω λοιπόν σε διάφορα σημεία αυτής της οδηγίας για τις διαδικασίες. Ζητούμε να υπάρχουν ε, κοινέ διαδικασίες και όχι κατώτατες προδιαγραφές βάσει του ότι ε, λέγουν οι ε, συνθήκες και αυτό πρέπει να τονιστεί. Επίσης πρέπει να βασιστούμε ή στην ομολογία του δικαστηρίου και να τονίσουμε ε, αυτό το οποίο ε, έχει λεχθεί σχετικά με την κατάρτιση των υπευθύνων ε, και ιδίως όσον αφορά τα ευάλωτα άτομα και τα άτομα που έχουν βασανιστεί και συγχρόνως να εντοπίσουμε τις ειδικέ ανάγκες και πάντοτε αναφερόμενοι στη σχετική οδηγία. Σας ε, αναφέρω αυτά τα σημεία για να σας πω τι πάει καλά και ε, το άλλο το οποίο ίσως δεν αντιμετωπίσαμε με τον ίδιο τρόπο και αναφέρω εδώ ως σημείο ανικανοποίησης ε, δύο στοιχεία. Καταρχήν ε, η ευελιξία των <clears throat> θεμάτων όταν ένα κράτος ε, έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα συγχρόνως πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αυτή την πίεση και ε, τον υψηλό αριθμό ατόμων που ζητούν προστασία και αυτό αναφέρεται στα άρθρα και πολλές φορές δεν υπάρχει μόνο ο προστα... Ε, ε, ε, δεν χρειάζεται μόνο προστασία αλλά ίσως χρειάζεται και υπέρμετρη υπάρχει υπέρμετρη πίεση για να υπάρξει αυτή η προστασία και πρέπει να επιτύχουμε ε, μεθόδους ε, εθνικές ε, που είναι διαφορετικές και να μπορέσουμε να τις ενοποιήσουμε. Να υπάρξει ευρέως ο σεβασμός της προθεσμίας του εξαμήνου για την απόδοση μίας αποφάσεως διότι υπάρχει μία κατάσταση σε διάφορες χώρες η οποία είναι προσωρινή και μπορούν με αυτή τη στιγμή να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που εψέρχονται σε αυτή την κατηγορία, υπάρχουν πολλά σημεία ασάφειας ε, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να υπάρξουν πολλές επιπτώσεις. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μάλλον Ήθελα να βραχυνθούν οι προθεσμίες. Ε, είναι ορισμένα σημεία επί των οποίων θα συνεχίσουμε να συζητάμε και όσον αφορά τη διαδικασία θέλω να καταλήξω διότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα όσον αφορά ε, αυτή την οδηγία για τις διαδικασίες. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη χαιρέτησαν την προσπάθεια ε, και ε, έχουν ορισμένες ανησυχίες, αλλά έχει ανησυχίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει λοιπόν με την ευκαιρία αυτή να ακούσουμε πολύ σύντομα πού έχουμε κάποια πρόοδο και να καταφέρουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα να καταλήξουμε σε μία συμφωνία σχετικά με αυτή την οδηγία για τις διαδικασίες. Ε, σας ευχαριστώ. Όντως πολύ αποτελεσματικά καλύψατε το κενό και θεωρώ ότι είναι καλό τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την κυρία Γκάν η οποία θα μας δώσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μας την παρουσιάσει και μετά θα ακούσουμε τον ε, Πολωνό Υφυπουργό ο οποίος έφτασε ήδη. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Γκάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για να δώσω στην Προεδρία να ξεκινήσει τη συζήτηση με την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την επιβεβαίωση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναμορφώσει την πολιτική ασύλου και να την προσαρμόσει εις τις προτάσεις που θα καλύπτουν τους ετούντες άσυλο για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο που έχει τεθεί για το 2012. Χάρη στην γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ε, ε, περιασμένη άνοιξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπόρεσε να καταλήξει σε μία ισοσχελισμένη πρόταση μεταξύ αποτελεσματικότητος ε, και δικαιοσύνης του συστήματος και πολύ, πολύ προσεκτικά άκουσα τα σημεία που δεν ικανοποιούν το Κοινοβούλιο Όπω όπως είπε η συγγήτρια. Ε, πιστεύω όμως ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να κρατήσουμε μία ισορροπία σε αυτήν την ε, οδηγία και να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες τις οποίες ανέφεραν τα κράτη-μέλη κατά την ε, συζήτηση της ε, ε, πρώτης, του πρώτου κειμένου αυτής της διαδικασίας. Βλέπουμε ότι πολλές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ήδη μορφώσει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την δικαστική βοήθεια βοήθεια τη σύγχυση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων πρωτοδικίων και εφετείων είναι θέματα τα οποία λάβαμε υπόψη μας διότι εάν υπάρχουν ευάλωτα άτομα ή θέματα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επίσης πρέπει να σημειώνουμε τους λόγους που οδηγούν σε μία επιτάχυνση της διαδικασίας. Μία άλλη βασική τροπολογία την οποία δεν δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι τροπολογίες σχετικά με τις ασφαλείς χώρες διότι εμείς ε, αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου ότι δηλαδή δεν υπάρχει ακόμη εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου των Ασφαλών Χωρών αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή ακόμη και έπρεπε να αφήσουμε τη δυνατότητα στο γραφείο των χωρών ασύλου να προωθήσουν την κατάσταση ιδίω βάσει κοινών ε, εκθέσεων που θα πρέπει να καταρτιστούν. Όταν λοιπόν ε, θα υπάρχει ε, και θα έχει αποκρισταλωθεί η δυνατότητα ευρωπαϊκής αναλύσεως θα μπορέσουμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό σε μια περαιτέρω φάση εναρμονίσεως στην Ευρώπη και εντωμεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, επανεξετάζει τακτικά σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ε, το Συμβούλιο την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στα κράτη-μέλη. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά την αντίδραση αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε ε, εν ονόματι της Επιτροπής, ευχαριστούμε και την εισηγήτρια κυρία Γκυγιόμ και σας υπενθυμίζουμε ότι θα ξανασυζητηθεί αυτός ο φάκελος στις 11 ε, Οκτωβρίου. Θα υπάρχει δηλαδή επαρκής χρόνος για να το ξανασυζητήσουμε. Και τώρα έχουμε τον ε, Γενικό Γραμματέα, υφυπουργό του, ο, της Πολωνίας, ε, ο οποίος εκπροσωπεί τον Υπουργό κύριο Μίλλερ ο οποίος έρχεται κατευθείαν από το ΦΥΡΟΜ από τη συζήτηση που έγινε εκεί ε, και ε, παρουσίασε την έκθεσή του επ' αυτού εις ε, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και τον χαιρετίζουμε που θα παρουσιάσει αυτό το θέμα εν ονόματι της Πολωνικής Φροεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εκ μέρου τη Πολωνική Προεδρία θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πώς έχει κατάσταση με το πακέτο ασύλου και να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα του δεύτερου τμήματος της Πολωνικής Προεδρίας. Το κοινό σύστημα ασύλου, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και η ολοκλήρωση των εργασιών σε αυτό το δεύτερο στάδιο αποτελεί η προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας. Και είναι μία από, τις, από τα στοιχήματα της Πολωνικής Προεδρίας. Όπως ξέρετε, αυτό το πακέτο ασύλου αποτελείται από πέντε προτάσεις, την οδηγία για τα προσόντα, είναι οδηγία αυτή που είναι πιο κοντά στην έγκριση, στην υιοθέτηση και αυτή η υιοθέτηση δεν εξαρτάται από τη συζήτηση για το περιεχόμενό της, ε, αλλά από το να μπορέσει ε, να, υπάρξει μια συμφωνία για τους πίνακες αντιστοιχίας. Ελπίζουμε να μπορέσει να εγκριθεί λοιπόν αυτή η οδηγία. Κατόπιν έχουμε τον κανονισμό του Δουβλίνου και εδώ η Πολωνική Προεδρία από την αρχή, από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης που έλεγε το στο ΣΟΠΟΤ φέτος τον Ιούλιο. Αναμένει μια λύση που να μπορέσει να εξελίξει τις εργασίες. Έχουμε συζητήσεις με την Κομισιόν αλλά και με τα κρατημέλη για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Θεωρούμε πως αν μετά από τη μεγάλη πάυση δεν ξεκινήσουν και πάλι οι συζητήσει για το έγγραφο αυτό υπό την Πολωνική Προεδρία, οι πιθανότητε να εγκριθεί το έγγραφο αυτό μέχρι το τέλο του έτου θα είναι πάρα πολύ μικρέ. Μετά, το επίσημο, μετά το επίσημο συμβούλιο που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο, όπου τέθηκαν ερωτήσεις στους υπουργού σχετικά με τους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το έγγραφο, δηλαδή το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης ε, και ενημέρωση σχετικά με τις απειλές που θα μπορούσαν να υπάρξουν σε μια συγκεκριμένη χώρα σε σχέση με το σύστημα ασύλου και συγκεκριμένα η έλλειψη προετοιμασίας ενός, ε, μάλλον κάποιων κρατών μελών για να λάβουν ένα μεγάλο αριθμό ετούντων άσυλο και να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με όλες ε, τις μεταφορές. Μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι υπουργοί ενέκριναν ε, τον πρώτο μηχανισμό, αλλά δεν συμφωνούσε η πλειοψηφία σε σχέση με το δεύτερο μηχανισμό. Σε ορισμένες από τις παρεμβάσεις δινόταν ε, η δυνατότητα να υπάρχει ένα σύστημα που να λαμβάνει ως βάση, ως βάση τον ε, κανονισμό του Δουβλίνου ή άλλα νομοθετήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεδρίασης, η Προεδρία προετοίμασε ένα άλλο συμβιβαστικό παροετοιμασε ενα όπου συμπεριλαμβάνονταν ε, διάφορες προτάσεις συμβιβασμού και ελπίζω αυτή την εβδομάδα να μπορεί να στελεί το έγγραφο στο κρατη αν ε, τελικά το έγγραφο αυτό σταλεί στα κράτη-μέλη, το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων ε, θα διαβιβαστεί μέσω του Υπουργού Μίλλερ και στη συνεδρίαση που θα γίνει ε, στις Οκτωβρίου και μπορώ να σας πω ότι προχωρούμε και με τις προτάσεις οδηγίας που παρουσιάστηκαν την 1η Ιουνίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορώ να σας πω εγώ ότι στην Προεδρία έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχει αναλάβει την παρακολούθηση αυτών των ε, νομοθετημάτων και ελπίζουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο στις συζητήσεις μας κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας σε ό,τι αφορά την οδηγία σχετικά με την υποδοχή. Στην πρώτη ομάδα εργασίας ε, κατορθώσαμε ήδη να πετύχουμε ένα συμβιβασμό στη, και εγώ θα έλεγα ότι η πρόταση, την πρόταση αυτή την υποδέχτηκαν θετικά τα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι τις επόμενες συνεδριάσεις ε, που θα λάβουν χώρα για την οδηγία αυτή και συγκεκριμένα μετά τη συνεδρίαση της ΣΚΙΦΑ που θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο, ελπίζουμε να μπορούν να συμπεριληφθούν πιο πολιτικά παρά τεχνικά στοιχεία και στην ομάδα ΣΥΛΟΥ που θα λάβει χώρα στις 19 Οκτωβρίου ελπίζουμε να μπορέσει να διευκρινιστεί και ποιο είναι το πανόραμα σε σχέση με τις προσδοκίες των κρατών μελών για ποια σημεία μπορεί να συμφωνήσει η Κομισιόν και πού μπορούμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά αυτή την οδηγία σε σχέση με τις υποδοχές. Και ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας να μπορέσει να σημειωθεί και πρόοδος με αυτό το θέμα σε σχέση τώρα με την οδηγία για τις διαδικασίες. Έγιναν τέσσερις συνεδριάσεις της ομάδας ασύλου επικεντρώθηκαν ε, κυρίως ε, επί των ίδιων θεμάτων, δηλαδή στην πρώτη ανάγνωση της οδηγίας. Ξέρω ότι ακούστηκαν πάρα πολλές παρατηρήσεις ως προς ε, το περιεχόμενο και μπορώ να σας πω ότι έχουμε περίπου 100 επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της οδηγίας αυτής. Επίση μπορώ να σας πω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ανάγνωσης προετοιμάσουμε μια συμβιβαστική πρόταση που θα περιλαμβάνει αυτά τα στοιχεία τα οποία εμείς θεωρούμε ε, ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία. Αύριο θα λάβει χώρα νέα συνεδρίαση της ομάδας ασύλου όπου θα συζητηθούν αυτές οι συμβιβαστικές προτάσεις της Προεδρίας στη συνεδρίαση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τους υπουργού. Ο δικός μας υπουργό θα προσπαθήσει να αξιολογήσει τις ε, δυνατότητες συμβιβασμού προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μπορώ να σας πω ότι οι κύριες επιφυλάξεις ή τα σημεία στα οποία αναφέρθηκαν τα κράτη-μέλη είχαν να κάνουν ε, με τη ε, θέμα της κράτησης, το θέμα της επιταχυμένης διαδικασίας, ε, δηλαδή να δούμε πώς θα γίνει η μεταχείριση των μετέπειτα αιτήσεων και Επίσης, να μπορεί να επιληθεί και το πρόβλημα να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα προσφυγής. Αυτά ήταν τα κυρία κρεμή ζητήματα. Μπορώ να σας πω ότι εμείς ε, ήδη ανασκουμπωθήκαμε και αρχίζαμε να δουλεύουμε επί των εγγράφων αυτών μαζί με την ε, Προεδρία της Δανίας για να μπορεί να υπάρξει μια ρευστή συνέχιση στις συζητήσεις των, πακέλων, των φακέλων αυτών και επίσης συνεργαζόμαστε και με το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ομάδας επαφής ε, που δημιουργήθηκε στο ΣΟΠΟΤ με πρωτοβουλία της Προεδρίας και ελπίζουμε να μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των εργασιών για τα εγγραφευτά. Επίσης, ε, θέλαμε να σημειώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο επί την Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστώ. Thank you. On behalf of the Polish presidency for... Και εμείς σας ευχαριστούμε, εξ ευχαριστούμε την Πολωνική Προεδρία. We should get started back to Madame Guillaume pour commenter. Κυρία Γουλιέλ μου για να σχολιάσει. Ορίστε. Τρία σχόλια. Πρώτον αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, αυτό το ξέραμε. Καμιά φορά βέβαια η συγκυρία ως προς τους μετανάστες μας αναγκάζει να θεωρήσουμε ότι το άσυλο έχει όντως μια ιδιαιτερότητα, δεν πρέπει να το θεωρούμε ως συνονθήλευμα με άλλα θέματα. Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να συνεχιστούν οι εντάσεις, έστω και αν είναι προσωρινές, αλλά να υπάρξει ένα σύστημα ασύλου που να δίνει μια πραγματική και μόνιμη λύση και όχι απλώς ένα μπάλωμα για τα εθνικά συστήματα. Αυτά όλα είναι νομίζω σημαντικά. Δεύτερον, για τη δέσμη του ασύλου γενικότερα. Μας είπατε ποιες συζητήσει γίνονται, ποια είναι τα θετικά σημεία και ποια είναι τα αδύνατα. Είπε η Πολωνική Προεδρία ποιοι είναι οι μηχανισμοί έκτακτης μεταχείρισης. Υπάρχει αυτό το λεγόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και το σύστημα αξιολόγησης. Πρέπει όμως να μην καθιστούν τα πράγματα ακόμη δυσκολότερα και πιο πολύπλοκα αλλά να διασφαλίζουν κάποια ρευτότητα και συνέχεια για να μπορεί να εγκριθεί ως το δυνατόν πιο εναρμονισμένη λύση. και φυσικά με βάση τα πέντε κείμενα που αναφέραμε τέλος για το 2012 ευχαριστώ την Πολωνική Προεδρία που δέχτηκε να συζητήσει το θέμα για να υπάρξει κάποια πρόοδος και να προχωρήσει η διαπραγμάτευση με κάποιο στόχο όμως για να προοδεύσει και το περιεχόμενο. Εγώ και ελπίζω και το Κοινοβούλιο έχουμε στόχο να υπάρξει λύση με σεβασμό βέβαια τη θεσμική ισορροπία. Ευχαριστούμε. Φράου Χολμάγερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, ε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία η οποία κάνει ε, πολύ φιλότιμες προσπάθειες για να αποδεσμεύσει τα μπλοκαρισμένα θέματα και να τα οδηγήσει σε μία αίσια επίλυση κατά τρόπον ώστε στο τέλος να καταλύσουμε σε ένα εναρμονισμένο πακέτο ασύλου στην Ευρώπη. Όσον αφορά την οδηγία για την διαδικασία θεωρώ ότι είναι θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις νομικές συμβουλές βασίστηκε στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προσήγγισε και τις θέσεις των κρατών όταν υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια και για τις ιδιωτικές αιτήσει. Βλέπω βλέπω ότι υπήρξαν θετικές προσεγγίσεις των θέσεων από μέρους Επιτροπής ε, μαζί μας και επίσης όσον αφορά ε, την, ε, την ε, ε, σιωπηλή ε, αναπομπή των αιτήσεων οδήγησε τα κράτη-μέλη να αποδεχθούν τις θέσεις τις οποίες είχε προωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε όμως ορισμένα προβλήματα. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε μία γρήγορη και συνεκτική διαδικασία. Εάν αυτό το θέλουμε για να βοηθήσουμε τους πραγματικούς προσφυγές θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο πρόσφυγας να δώσει όσες αναγκαίες πληροφορίες χρειάζεται για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή η αίτησή του σαν πρόσφυγα εγκαίρος και ε, έτσι δεν θα έχουν πολλές δυνατότητες τα κράτη-μέλη για παρεκτροπές ή ε, ε, δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν με κακό σκοπό ορισμένοι το δικαίωμα αυτό ασύλου για να αποκτήσουν ταξιδιωτικά έγγραφα και διότι προσπαθούμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους διαδικασίες. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι ίσως προβληματικό σημαντικό όταν ε, ε, υπάρχει ε, αναγνώριση ενός δικαιώματος εισόδου υπάρχει αυτομάτως και ένα δικαίωμα παραμονής. Εάν όμως κάποιος προσπαθεί απλώς να πάρει μία παράτηση χωρίς να προσκομίζει νέα στοιχεία θα έπρεπε να μην υπάρχει υπάρχει αυτόματη ανανέωση της διαμονής και να εμποδιστεί μια τέτοια διαδικασία διότι πολλές χώρες έχουν διαπιστώσει ε, ατυχώς ότι υπήρξαν ε, πολλές εκμεταλλεύσεις ε, αυτών των δικαιωμάτων και υπάρχουν παρεκτροπές σε πολλά κράτη-μέλη χωρίς όμως να μπορεί κανείς να ε, εμποδίσει την κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για το σωστό σκοπό. Θέλουμε μια πιο γρήγορη μεν διαδικασία αλλά αυτό σημαίνει ότι αν υπάρχει κατάχρηση θα πρέπει να ανταδρούμε και πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή εάν υπάρχει μια ε, συμπληρωματική αίτηση θα πρέπει να ε, την ε, εξετάζουμε μαζί με την αρχική για να βοηθήσουμε τον πρόσφυγα. Εάν όμως καταφανώς πρόκειται για κατάχρηση των δικαιωμάτων θα πρέπει στη δεύτερη αίτηση ή στην τρίτη αίτηση να υπάρχει μία γρήγορη διακασία, πιο, ε, ε, με μεγαλύτερη επιτάχυνση δηλαδή, ιδίως ε, σε χώρες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλαπλές περιπτώσεις και έχουν και οικονομικές δυσκολίες. Καταλαβαίνω τα προβλήματά τους, αλλά γι' αυτό θα έπρεπε τουλάχιστον να συζητήσουμε, όπως και στο θέμα των επιταχυμένων διαδικασιών, την, την παραβίαση του δικαιώματος συμμετοχής. Εάν κάποιος δηλαδή ε, δεν συνεργαστεί, δεν συμπράξει, ε, θα πρέπει να ε, μην του ανοίξουμε την πόρτα να εφαρμόσει αυτές τις μεθόδους διότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος χωρίς έγγραφα ή με παραποιημένα έγγραφα έχει μεν ταξιδέψει και ε, κοιτάζει ε, να να ε, ε, ε, μπει σε μια χώρα. Εάν υπάρχουν έλεγχοι οι οποίοι αποδεικνύουν ότι σωστά έφτασε, έχει καλός. Αλλά όταν υπάρχει εσκεμένα ένα παραποιημένο όνομα, όταν υπάρχουν σαφώς πλαστά έγγραφα, τότε από την αρχή δεν πρέπει κανείς να προωθήσει σε μία διαδικασία παρατάσεως της, πα, της παραμονής. Αυτά όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να εξεταστούν και σε επίπεδο κρατών μελών και να τα επιλύσουμε όλοι μαζί. Όσον αφορά τις ειδικέ ανάγκες νομίζω ότι όπως ήδη ελέγχθη χρειαζόμαστε μεν διαδικασίες κατά, κατά περίπτωση αλλά δεν χρειάζεται να είναι αυτοματοποιημένη η μέθοδος που οδηγεί στην χορήγηση κάποιου καθεστώτος. Δηλαδή Δηλαδή ε, δεν, είναι δυνατόν κάποιος 26 χρονών επειδή ε, θεωρείται ότι έχει περάσει δύσκολα να έχει ειδικέ ανάγκες ε, που να τον διαφοροποιούν από κάποιον άλλον της ιδίας ειδικίας, διότι τελικά αυτό που πρέπει να προτεύσει στην περίπτωση αυτή είναι η συγκεκριμένη προσωπική του κατάσταση η οποία θα πρέπει να εξεταστεί καλύτερα και θα ήθελα να κάνω μία ακόμη πρόταση η οποία ε, μου έχει προταθεί από αυτούς οι οποίοι κάνουν τις συνεντεύξεις Δηλαδή οι ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι επιβαρύνουν τους υπευθύνου αυτούς για συνεντεύξεις. Ναι μεν χρειάζονται μία βοήθεια διότι έχουν δυσκολία να προσαρμόσουν τις συνεντεύξεις τους στις δικές μας ανάγκες διότι είναι υπερβολικά βεβαρημένοι. Χρειάζονται λοιπόν κάποιες συμβουλές αλλά ε, υπάρχει και το θέμα του Ιάσο το οποίο θα μπορεί να συνεργαστεί με διάφορες ε, άλλες οργανώσεις και να καταρτιστεί ένας ευρωπαϊκός κανόνας σχετικά με τις χώρες προελεύσεων ώστε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για το πώς θα αντιμετωπίσει κανείς και το Ιάσο. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης αλλά πριν η κυρία Βίξτρομ. Ε, ένα διαδικαστικό. Έχουμε, ε, ε, έχουμε απεριόριστο χρόνο ομιλίας, διότι στο τέλος θα καταλήξει ότι ορισμένοι από εμά θα έχουν 20 δευτερόλεπτα για να μιλήσουν και αυτό δεν είναι σωστό. Βεβαίως, ουσιαστικά ποτέ εδώ δεν υπάρχει άκρατος χρόνος ομιλίας και απεριόριστος. Το θέμα είναι ότι έχουμε προβλέψει ε, μία ε, ψηφοφορία στις 12. Οπότε έχουμε ακόμη περίπου 15 λεπτά, 10-15 λεπτά. Δέκα μάλλον λέει ο πρόεδρος αλλά ε, ε, υπάρχουν διάφοροι ε, ευρωβουλευτές που θέλουν να παρέμβουν και εσείς κυρία Βίξτρομ και προσπαθούμε πάντοτε να είμαστε ευέλικτοι το έχετε διαπιστώσει πάντοτε οπότε σεβόμαστε όλους αυτούς που θέλουν να μιλήσουν αλλά επίσης πρέπει να υπάρχει και αυτοπεριορισμός γνωρίζοντας ποιο είναι το πρόγραμμα της Επιτροπής η κυρία Γκυγιόμ Συγγνώμη. Ε, μίλησα για ένα συγκεκριμένο θέμα και ένα συγκεκριμένο κείμενο που ήταν στην εμπειρία διάταξη. Μου φάνηκε τώρα ότι μιλάμε γενικά και ήμασταν εδώ για να ακούσουμε τον κύριο Υφυπουργό για το πακέτο ασύλου στο σύνολό του. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μια τέτοια συζήτηση χωρίς να μπαίνουμε ε, σε πάρα πολλές λεπτομέρειες επί του ενός κειμένου. Αυτό κατάλαβα, κάνω λάθος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Υπουργό έχει σημειώσει τα σχόλια, αλλά θα ακούσουμε. Έχω τρία μέλη. Πριν να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Υπουργό και βλέπετε την κυρία Κέλλερ. Θέλετε να πάρετε το λόγο, μάλιστα. Τέσσερις. Ο κύριος Τριδεφιλίδης. Και προτείνω να περιοριστείτε στα χρονικά όρια, γιατί έχουμε και την ψηφοφορία στις 12. No chairman. Μη φοβάστε, Πρόεδρε. Ένα λεπτό μόνο και τρία δευτερόλεπτα. Θα περιοριστώ σε ένα σχόλιο που έκανε η Προεδρία. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Προεδρία για την περιγραφή της κατάστασης σε ό,τι αφορά την οδηγία περί προσόντων, τον κανονισμό του Βλήνου, την οδηγία για τις διαδικασίες υποδοχής. Αλλά θέλω να σταθώ σε ένα θέμα που αφορά το μηχανισμό αξιολόγηση και το σύστημα εγκαίρη προειδοποίηση. Φαίνεται να προτείνει η Προεδρία ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο κανονισμό του Δουβλίνου, ενώ πιστεύω ότι είναι λάθο. Θα προτιμούσα αυτό να βρίσκονται σε όλες τις οδηγίες, κυρίως ό,τι αφορά τις οδηγίες περί διαδικασίας, τη οδηγία περί υποδοχής. Χρειαζόμαστε εκεί κάτι τέτοιο περισσότερο παρά τους κανονισμούς του Δουβλίνου, όπου φυσικά το κρεμίσταμα είναι ε, να σταματήσουν ε, οι μεταφορές. Μάλιστα, πολύ καλά. Η κυρία Φαγιόν. Ehm, Ευχαριστώ. Θέλω να αντράξω την ευκαιρία, καθώς έχουμε εδώ τον κύριο Φιπουργό που μόλις ήρθε από την Οχρίδα, που εξακολουθούν μιλάνε, να μιλάνε για τις διαδικασίες πλαστών, πλαστοποίησης θεωρήσεων. Αυτό έχει συμβεί τελευταία πολλές φορές ε, στο Βέλγιο και στα κανονικά κράτη. Βρήκαμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους ε, από τη Βασιλεία Τσεκοβίνη, ετούντες άσυλο. Και το τονίζω αυτό για να σας πω γιατί χρειαζόμαστε τις καταλληλές διαδικασίες ασύλου. Τι συμβαίνει, οι πολίτες αυτοί εκμεταλλεύονται πιο ευνοϊκές διαδικασίες ασύλου ε, λαμβάνουν ε, καλύτερες ε, προϋποθέσεις υποδοχής και θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε φτάσει σε κάποιες βαρχιπρόθεσμες αποφάσεις σε σχέση με το πώς ε, θα αντιδράσετε για να αποφύγουμε αυτές τις ψευδείς αιτήσει. Και θα ήταν δυνατό να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα στο σύνορο με την Ουγγαρία για να παρεμποδίσουμε την εισρωή νέων μεταναστών από τα Βαλκάνια καθώς και μετανάστες που περνούν από το σε αυτό και έρχονται από τον αραβικό κόσμο. Κύριε Δίκστρομ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία Δεν μπορούμε να θεωρούμε την Πολωνία ως νέο κράτος μέλος πλέον, αλλά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Εσείς ε, προωθήσατε το φάκελο του ασύλου, το εκτιμούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάλι σας ευχαριστούμε. Επίσης, ε, οι πρωτοβουλία δημιουργίας μιας ομάδας εργασίας. Και εμείς ε, θέλουμε να συνεισφέρουμε σε αυτό στο μέτρο του δυνατού. Θα είμαι σύντομη. για την οδηγία των προσόντων. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα σε συμφωνία και ελπίζω ότι η οδηγία για την υποδοχή και η οδηγία για τις διαδικασίες ε, να ε, καταλήξουν κάπου, επιτρέποντας έτσι να ανοίξει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Είμαι συγγήτρια για τον κανονισμό αυτό και παρακολουθώ την ε, εμπλοκή στο Συμβούλιο και πραγματικά εκτιμώ τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε καθώς και τη βούλησή σας να βρεθεί μια κοινή λύση. έτσι ώστε να μην ε, ισχύσει ο εθνικισμός. Μάλιστα. Κυρία Κέλλερ, εδώ δεν συζητάμε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου καθεαυτές. Η Πολωνική Προεδρία υποτίθεται ότι θα μας έκανε μία πρόταση συμβιβασμού. Δυστυχώς δεν άκουσα καμία τέτοια. Μας παρουσιάσατε ένα χρονοδιάγραμμα, πότε θα συνεδριάσει η ομάδα εργασίας για το άσυλο κτλ. Αλλά ποιος είναι ο συμβιβασμός. Αυτό θέλουμε να μάθουμε, αφού θέλουμε να γνωμοδοτήσουμε. Ίσως μπορείτε να μας πείτε λοιπόν. Ο κύριος Μπουζούτιλ. για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Στις 22 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δύο εβδομάδες περίπου πριν, ο Γενικός εισαγγελέα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέβαλε μία γνωμοδότηση όπου έλεγε ρητά ότι δεν πρέπει μια χώρα να ξαναστέλνει πίσω στη χώρα προέλευσης του έναν αιτητή ασύλου εφόσον υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μπορεί εκεί να παραβιαστούν τα ανθρώπινά του δικαιώματα. Έχουν όμως σταλεί άνθρωποι από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα πίσω και ο Γενικός Αγγελεύς λέει ότι αυτό το εξής πρέπει να απαγορεύεται. Το Συμβούλιο όμως δεν απαντάει σε μία πρόταση της Κομισιόν από το Σεπτέμβριο του 2008 σχετικό, σχεδόν τρία χρόνια πριν. και ακόμη το Συμβούλιο δεν έχει νομοθετήσει. Η, τα αποτελέσματα είναι σαφή. Αφήνουμε το δικαστήριο να αποφασίζει για την νομοθεσία αντί να νομοθετούμε εμείς. Και μας λένε συνεχώς ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει ως έχει. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Υπουργό το Συμβούλιο προτίθεται ή όχι να κάνει οποιονδήποτε συμβιβασμό για αυτή την πρόταση. Ευχαριστούμε. Ο Υφυπουργό έχει σίγουρα σημειώσει, ο Υπουργό μας έχει σημειώσει τις παρατηρήσεις αυτές. για τη δέσμη του ασύλου. Έχει δοθεί μια νέα όθηση γιατί έχει προσέξει το θέμα ιδιαίτερα η Πολωνική Προεδρία και θα μας απαντήσει στον τελευταίο γύρο. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Φυσικά τα λαμβάνουμε θα τα λάβουμε υπόψη μας όταν συντάξουμε τις προτάσεις της Προεδρίας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι βλέπετε όπως και εγώ ότι τα έγγραφα που αφορούν το άσυλο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συνταχθούν εφόσον θέλουμε να εξισορροπήσουμε το σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτητών. Απ' την άλλη δε τα αιτήματα των χωρών μελών που θέλουν να αποτρέψουν τη χορήγηση ασύλου σε όσους τη ζητούν ε, αθέμητα. Υπάρχουν οι πραγματικοί αιτητές ασύλου και ορισμένοι άλλοι που το χρησιμοποιούν ως πρόφαση. Όσοι πράγματι χρειάζονται βοήθεια πρέπει να μπορούν να τη λαμβάνουν πολύ πιο σύντομα από ό,τι μέχρι τώρα. Μπορεί όμως να υπάρχει και απειλή για την ασφάλεια μιας χώρας εάν υπάρχει κατάχρηση του συστήματος. Και αυτά σχετίζονται και με την πολιτική των θεωρήσεων και την προστασία των συνόρων. Αυτά που διαπίστωσα εγώ είναι ότι η εξισορρόπηση αυτών των δύο είναι το σημαντικότερο θέμα εδώ για το άσυλο. Όσο για το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, θα θέλαμε να μην είναι δημο... Ε, γραφειοκρατικός αλλά να αντιδρά με βάση τα στοιχεία που θα μας έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να μας επιτρέπει να δούμε σαφώς ποιες χώρες μέλη είναι έτοιμες, διατεθειμένες να δεχτούν πρόσφυγες και ποιες όχι αυτές που δεν είναι σε θέση να τους δεχτούν θα έπρεπε να τύχουν της βοήθειας κάποιων μηχανισμών που υπάρχουν μεν αλλά ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουν να τους χρησιμοποιήσουν όπως πρέπει. Σε επίγουσες καταστάσεις δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θεωρούμε. Για το Δουβλίνο καταλαβαίνω ποια είναι η κατάσταση και νομίζω ότι μετά από την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου υπήρξε συμβιβασμός Γνωρίζουμε το εύρος του, γνωρίζουμε τι μπορούν να δεχτούν οι χώρες μέλη και τι δεν μπορούν. Και αυτό ακριβώς το θέμα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε σαφέστερα Το σύστημα που προτείνουμε προβλέπει την αξιολόγηση και των πληροφοριών από τις χώρες μέλη και την υποβοήθησή τους ώστε στο μέλλον να μην υπάρχει καμία χώρα μέλος όπου ένας αιτητής ασύλου να χρειάζεται να μεταφερθεί κάπου αλλού γιατί δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες διαβίωσης του. Εχθές έγινε μια πολύ ζωηρή συζήτηση μεταξύ Προεδρίας και Κομισιόν με εκπροσώπους Βαλκανικών κρατών. Και νομίζω ότι όλοι συμφώνησαν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να περιοριστεί το φαινόμενο της κατάχρησης του συστήματος του ασύλου. Τώρα οι συμβιβασμοί και τι προτείνουμε για την οδηγία υποδοχής τι προτείνουμε για το Λουβλίνο σας είπα ότι και τα δύο αυτά θέματα θα σας υποβληθούν από τον Υπουργό Μίλερ στις 12 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας Και τώρα παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνεται μία εκδήλωση για το άσυλο από τον συνάδελφο Κλωτ Μωράες με τον Ερυθρό Σταυρό, τα Ηνωμένα Έθνη, το Ινεπάτη Αρμοστία για τους πρόσφυγες μία συζήτηση και μία φωτογραφική έκθεση για τους αιτητές ασύλου στην Ένωση. Θα οργανωθεί στο κτίριο Αλτιέρου Σπινέλη στις 6 το απόγευμα στις 18 η ώρα. Ευχαριστούμε τον Υπουργό λοιπόν και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών όπου θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Καθίστε παρακαλώ και ετοιμαστείτε για την ψηφοφορία. I can promise that we will make what will be possible. Thank you. Thank you. Bye.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 Dear colleagues, if you're all ready, not to have complaints about the timing, please. Αν είστε έτοιμοι συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση των Επιτροπών Λίμπη Λοιπόν, όπως είχε προγραμματιστεί, έχουμε και τη συνεδρίαση των δύο Επιτροπών και Καταρχήν να συγχαρούμε τον συνάδελφο, τον κύριο Μάικλ Κούσταυσον, οποίο είναι ο αναδιοριστέντας πρόεδρος της Επιτροπής ΦΑΜ. Ε, είχαμε ιδιαίτερα καρποφόρη συνεργασία με την Επιτροπή αυτή, τον καλωσορίζουμε και τον συγχαίρουμε για τα καθήκοντα που θα αναλάβει για την ανάληψη της Προεδρίας και θα του δώσουμε το λόγο να μας κάνει μια παρουσίαση. Uh, θα μιλήσω σουηδικά, δεν θα μιλήσω αγγλικά. Ναι, πραγματικά είμαι ολοκένουριος ως πρόεδρος. Χθε εξελέγει. Και για μένα είναι πραγματικά μια τιμή να αναλαμβάνω εδώ καθήκοντα τέτοιου είδου στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί στον ίδιο τομέα έχω εργαστεί και στη Σουηδία. Ως ε, πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών, να σας πω ότι το πρώτο μου καθήκον είναι να συμπροεδρεύσω σε αυτή τη συνεδρίαση μαζί σας, ε, κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η ψηφοφορία για την Ευρωπαϊκή Εντελή Προστασίας ε, είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί αυτό δείχνει ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη βία κατά των γυναικών. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, βεβαίω, ε, Πάρα πολύ σοβαρά λαμβάνουμε το θέμα που διακυβαίνεται εδώ, κυρία Λούτφορτ. Ευχαριστώ να καλωσορίσω ότι έχουμε έναν άντρα πρόεδρο της Επιτροπής ε, για τις Γυναίκες. Εγώ είμαι φεμινίστρια και με ενδιαφέρει ισότητα των γυναικών. Αλλά ανησυχώ ορισμένε φορές, ποτέ δεν ήμουν μέλος, το παραδέχομαι. Αλλά μήπω είναι πάρα πολύ περιορισμένη στον εαυτό τη ε, αυτή η Επιτροπή. Και όσοι υπόθηκαν μόλι, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Χρειαζόμαστε την ισότητα των γυναικών, ε, αλλά και την ισότητα ε, των ανδρών. Ε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε λοιπόν να ανοίξετε το θέμα αυτό. Δηλαδή να το εντάξετε σε ένα πλαίσιο σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου θα αφορά όλους. Ε, ελπίζουμε να πετύχετε και την πλειοψηφία αυτού του κοινοβουλίου και να μην υπάρχουν μόνο συζητήσεις. Αν τα καταφέρετε αυτά νομίζω ότι θα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, δεν είναι τώρα η ώρα να ανοίξουμε τέτοια συζήτηση σε σχέση με την ισότητα ανδρών και γυναικών. Αλλά ο κύριος Γκούστευσον φυσικά θέλει να αντιδράσει. Ε, eh, eh, ναι, δεν ξέρω τι έγινε στο παρελθόν, ε, πώς γινόταν ε, τα πράγματα στο παρελθόν, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι το θέμα ε, της ισότητας ε, των γυναικών, των δύο φίλων δεν είναι μόνο ένα θέμα που αφορά ε, τις γυναίκες μόνο, είναι ένα θέμα που αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει να συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο στην κοινωνία, να μην υπάρχουν διακρίσεις και βεβαίως και εγώ ως άνδρας υπερασπίζω αυτές τις αρχές γιατί με ενδιαφέρει, έχω ενδιαφέρον να υπερασπίσω αυτές τις αρχές. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον κύριο Γκούσταυσον. Τώρα, πρέπει να βάλουμε τελεία σε μια μακρά συζήτηση για αυτή την Ευρωπαϊκή Έντολη Προστασία. Καταναλώσαμε πολύ χρόνο και ενέργεια στις συζητήσεις μας και στις δύο επιτροπές, ε, και στην Επιτροπή Λίβη και στην Επιτροπή ΦΕΜ και υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, όμως τις ξεπεράσαμε με επιτυχία. Χάρη στη δουλειά που έγινε και από την κυρία Ρομέρο και από την κυρία Παχαιχαρίλη, από τις δύο και φυσικά από όλους τους κοιόδης και όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν. Και Επίσης και από κάποιο άτομο που, μας, που παρευρίσκεται εδώ, ο κύριος Περίλο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας που βοήθησε την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την εργασία της στο θέμα αυτό. Μας βοήθησε και πρόσφατα διορίστηκε και δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστούμε, λοιπόν. Ευχόμαστε... Σας ευχόμαστε. Καλή επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ. Λοιπόν, ίσως ε, οι συγγήτριες, ε, αν θέλουν να πάρουν το λόγο, οι συγγητές. Θέλετε να πείτε κάτι πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ. Κύριε Ρομέρο, ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε. Ναι, θέλω να πω κάτι, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τις ε, γυναίκες στην Ευρώπη, για τις Ευρωπαίες και είναι μια μεγάλη μέρα για την οικοδόμηση αυτού του χώρου δικαιοσύνη που θέλουμε για την Ευρώπη. Όχι μόνο μιλάμε για χώρο δικαιοσύνη, γιατί έχουμε δει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα αλλά πρόκειται και για ένα χώρο δικαιοσύνη. και γι' αυτό το λόγο το γεγονό να μπορούμε να έχουμε μια εντολή προστασία για όλα τα θύματα κυρίως για τις γυναίκες, αλλά όχι μόνο, αλλά και για τους ενηλίκους ε, και για όλες τις ε, ομάδες που υφίστανται επίθεση και που βρίσκονται σε κίνδυνο και θίγεται η κυριότητά τους. Ε, μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή σήμερα αυτό το μηχανισμό και μας φαίνεται ότι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα για την Ευρώπη. Γι' αυτό θέλω να το γιορτάσω και θέλω να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία που στις αρχές του 2010 ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, την κατέθεσε επιτάπητος και επίσης ε, τα κρατη που τη βοήθησαν, τα δύο κράτη-μέλη που τη βοήθησαν σε αυτή την πρωτοβουλία και σήμερα και την Πολωνική Προεδρία, γιατί χάρη στην Πολωνική Προεδρία κατορθώσαμε να απεμπλοκάρουμε τη διαδικασία και κατορθώσαμε αυτή η εντολή προστασία τελικά να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι το τελευταίο εμπόδιο το ξεπεράσαμε χάρη στην Πολωνική Προεδρία γιατί αυτή η εντολή προστασίας θα μπορούσε να αναβληθεί μέχρι ε, ο κανονισμός ε, που κατέθεσε η Κομισιόν να συζητηθεί. Ε, η όμως η Πολωνική Προεδρία κατόρθωσε να γίνει η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας μια πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν σήμερα κατορθώσαμε κάτι τέτοιο να αποτελεί ε, έκτακτη ανάγκη, δηλαδή ε, χάρη σε αυτή την απόφαση της Πολωνικής Προεδρίας, ακόμη και να γλιτώσουμε ένα θάνατο, τότε μπορούμε να πούμε ότι τα καταφέραμε. Ευχαριστώ η συνάδελφος που ήταν η για την Επιτροπή ΦΑΜ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουν ε, την Ευρωπαϊκή Εντήλη Προστασίας. Ε, ήταν δύσκολος ο δρόμος να φτάσουμε μέχρι εδώ, αλλά είναι μεγάλη μέρα σήμερα για όλους εμάς ε, και μπορούμε να αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη δουλειά που κάναμε. Πιστεύω ότι σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τα θύματα, για όλα τα θύματα. Ξέρουμε ότι αυτή η εντολή θα αποφελήσει κυρίως ε, τις γυναίκες, ε, όπως ε, η εντολή της απομάκρυσης που υπάρχει ήδη στη χώρα τους, θα μπορεί να εφαρμόζεται, να εκτελείται και σε άλλες χώρες. Αλλά η ιδέα αυτής της εντολής προστασίας γεννήθηκε για να καλύπτει και όλες τις ομάδες δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους ε, ανηλίκους, τα θύματα της τρομοκρατίας και οποιοδήποτε θύμα, άνδρα ή γυναίκα που αισθάνεται ότι είναι υποδιωγμό και θέλει να υποφελείται από ένα χώρο ασφαλείας. Εμείς ε, τι κάνουμε, αρχίζουμε τώρα να μεθυτούμε επί των θυμάτων. Από τη στιγμή που έφτασα εδώ, σε αυτό το κοινοβούλιο, είδα ότι υπήρχε μεγάλη έλλειψη για την νομοθεσία σχετικά με τα θύματα. Τώρα, χάρη στην Κομισιόν που παρουσίασε ένα πακέτο μια δεσμή μέτρων για τα θύματα, επί των οποίων θα είμαι και συγγήτρια, θα αρχίσουμε να αποδίδουμε δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια στα θύματα που αυτό ζητούν και το αξίζουν. Ευχαριστώ λοιπόν την Πολωνική Προεδρία που κατόρθωσε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια. Θέλω να ευχαριστήσω την Γραμματεία, ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια. Κάναμε πολύ καλή δουλειά πιστεύω και ευχαριστώ και όλους ε, τους κοιόδης εισηγητές. Και μπορώ να πω ότι σήμερα όλοι εμείς μπορούμε να είμαστε περήφανοι γιατί βοηθούμε όλα τα θύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλου του κόσμου γιατί θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ. Όπως ελέγχθη, είναι πολύ, ουσιαστικό, πολύ ουσιαστική κατάληξη για αυτό το βασικό θέμα το οποίο θέλει να συμβάλλει στο χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφαλείας. Να <clears throat> συμπληρώσουμε τις ευρωπαϊκές διατάξεις και να στείλουμε το μήνυμα προς Ευρωπαίους πολίτες ότι ενδιαφερόμαστε για αυτούς, για τα δικαιώματά τους, ε, ε, για την προστασία που τους οφείλουμε και ότι ε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να τους προστατεύσουμε με αυτή τη βασική πρωτοβουλία που ξεκίνησε με την Ισπανική Προεδρία και θα ψηφιστεί τώρα τελεσίδικα. Οπότε ψηφοφορία. Θέλετε ηλεκτρονική, θέλετε διατα... διανατάσεως χειρός ή έλεγχος ηλεκτρονικός. Νομίζω ότι ο έλεγχος θα μας δείξει πού πάμε. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγοι. Νομίζω ότι αυτό ήταν εξαιρετικό. 55 επί, ε, υπέρ, κανείς κατά και ευχαριστούμε τον κύριο Γκούσταυσον και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η εργασία με την Επιτροπή Γυναικών.